Αγαπητοί συνάδελφοι, γυναίκες από ό,τι βλέπω κυρίως, σας καλωσορίσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κατρίνα Σεσλέν Λανέλ, εκτελεστική διευθύντρια της ΕΦΣΑ. Ξέρετε ότι ήθιστε εδώ να βρισκόμαστε με την ΕΦΣΑ κάθε τόσο και να ανταλλάσσουμε απόψεις, απόψεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία δηλαδή Ασφάλειας Τροφίμων. Σίγουρα ο οργανισμός αυτός έχει έναν ανεξάρτητο και πολύ σημαντικό ρόλο και συγκεντρώνει πάρα πολλές γνώσεις και ξέρω τι λέω γιατί στην εκλογική μου περιφέρεια είχαμε σοβαρά προβλήματα κάποια στιγμή και η Εύσα μας βοήθησε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα και εντόπισε το πρόβλημα, αλλά και μας βοήθησε να το λύσουμε. Βέβαια, η κοινή γνώμη δεν τα γνωρίζει όλα αυτά. Εξάλλου, νομίζω ακριβώς γι' αυτό ότι θα πρέπει να φροντίσετε να προβάλλετε προς την κοινή γνώμη αυτά που κάνετε. Κατρίν, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα και που έτσι μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας. Συνεπώς, σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τόσο έχετε να μας πείτε και μετά θα έχουμε και συζήτηση φυσικά. Παρακαλώ, Κατρίν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Κρότε, αξιότιμα Ευρωβουλευτές. Σας είμαι ευγνώμων που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ετήσια πρόοδο της ΕΦΣΑ. Ξέρετε ότι η στήριξή σας στη δουλειά μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ήταν μεγάλη χαρά για μας επίσης που υποδεχτήκαμε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΕΝΒΗ υπό τον κύριο Χρότε στη Μπάρμα το Μάιο και έτσι σας δόθηκε ευκαιρία να δείτε πώς δουλεύουμε και τα δικά σας λόγια αποτέλεσαν ε, νέα έμπνευση για μας. Οι επαφές μας αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την υπηρεσία μας και για τη συμπίπτει με τη δέκατη επέτειο από τότε που άρχισε να λειτουργεί η ΕΦΣΑ, αλλά επειδή έχουμε και την ε, δημοσίευση της δεύτερης εξωτερικής αξιολόγησης της ΕΦΣΑ, κάτι το οποίο έχει επιπτώσεις για τις μελλοντικέ εξελίξεις στον οργανισμό αυτό και έτσι πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε την έκθεση αυτή μαζί. Οι απόψεις σας είναι ζωτική σημασίας προκειμένου να γίνουν συστάσεις που μας βοηθούν και προκειμένου να δοθεί και ένα κατευθυντήρια γραμμή στην ΕΦΣΑ. Μαζί με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ οργανώσουμε μία διάσκεψη ψηλού επίπεδου στις 13 Νοεμβρίου όπου η εξολόγηση αυτή θα έχει κέρια θέση στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζω να έρθετε όσο γίνεται περισσότερο από εσά στην Πάρμα. Οι διατάξει όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση της ΕΦΣΑ αναφέρονται στον ιδρυτικό μας κανονισμό, ο οποίος λέει ότι πρέπει να γίνεται εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού κάθε έξι χρόνια. Οι όροι της ε, δεύτερη αυτής αξιολόγησης αποφασίζονται ανάμεσα στην Κομισιόν και το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΦΣΑ. Η αξιολόγηση έγινε για ένα δωδεκάμινο από την Έρστεν Young μετά από έναν διαγωνισμό. Ένα μεγάλο μέρος ε, ενδιαφερομένων, ευρωβουλευτές, χώρες μέλη, επιτροπή, βιομηχανία με κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις καταναλωτών, ε, ερωτήθηκαν ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για όλες τις πτυχές της ΕΦΣΑ, την απόδοσή της, με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την απόδοση και την πρόσθετη αξία παρατηρήθηκε Μάλλον ε, παρατήρησαν, ήρθαν παρατηρητές και σε διάφορες συναντήσεις της ΕΦΣΑ και παρακολούθησαν και δραστηριότητές μας ε, σε συνδυασμό με άλλους ε, οργανισμούς διεθνείς ή σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ετοιμάστηκε και ένα έγγραφο με την ανάλυση της μελέτης αυτής. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής, ξεκινήσαμε τις διαβουλεύσεις μαζί σας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα κράτη-μέλη, με το Συμβουλευτικό Φόρου της ΕΦΣΑ, με την Επιστημονική μας Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε συστάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν αυτό ακριβώς το feedback. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι η ΕΦΣΑ λειτουργεί καλά, υποφέρει ε, καρπού ε, σύμφωνα με την αποστολή της και σύμφωνα με τις αξίες που υποστηρίζει. Φυσικά και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Είναι πάντω ενθαρρυντικό για όλους όσους συνεισφέρουν στο έργο μα να ακούμε απ' έξω από κάποιον ανεξάρτητο παράγοντα ποιε είναι οι συνέπειες, οι επιπτώσεις από το έργο του οργανισμού μα, που δίνει πολύτιμες από ό,τι φαίνεται επιστημονικές συμβουλές. Η έκθεση λέει ότι η ΕΦΣΑ συνεισφέρει στην ασφάλεια τρομίων στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρεται στην δυνατότητα της ΕΦΣΑ να συλλέγει επιστημονικές συμβουλές και πραγματογνωμοσύνη από το προσωπικό της, από διάφορα πάνελς, από εθνικούς εμπειρογνώμονες για θέματα ιδιαίτερα περίπλοκα και να μπορεί να ασχολείται πολύ καλά με την αξιολόγηση κινδύνων και με σχετικές ε, μεθοδολογίες σε όλο και περισσότερους καινούριου τομείς. Φυσικά χρειάζεται μεγάλη διαφάνεια και πολύ καλή οργάνωση για να τα φέρουμε σε πέρας. Αναγνωρίζει επίσης η έκθεση τη δουλειά που γίνεται με τους διάφορους ενδιαφερόμενους και ότι χρησιμοποιούνται επίσης πολλά μέσα για να πετύχουμε το στόχο μας. Επίσης μιλάει για την πρωτοβουλία μας να αναλάβουμε νέα βήματα για να κάνουμε αξιολόγηση κινδύνου. Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των ανακοινώσεών μας όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου αναγνωρίζονται, όπως επίσης και η συνεισφορά της ΕΦΣΑ για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι στα τρόφιμα που παράγει η Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι ολοφάνερο κυρίως στη συλλογή δεδομένων, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να πετύχει η αξιολόγηση κινδύνου. Και εξαρτάται βέβαια από τη συνεργασία των χωρών μελών. Η Ευρώπη έχει κάνει τεράστια βήματα σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Και η Επιτροπή αλλά και σε εθνικό επίπεδο όσοι ασχολούνται με την αξιολόγηση κινδύνου αναγνωρίζουν ότι έχουν στην διάθεσή τους πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά στοιχεία από εμά που βοηθούν στην αξιολόγηση κινδύνου για θέματα υγείας, για την ε, μικροβιολογική αντίσταση, ε, διοξίνες, παριστοκτόνα κτλ. Το βασικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι η επιστήμη είναι κεντρική σημασίας. Ξέρω ότι έχουν εκφραστεί πολλές ε, ανησυχίες όσον αφορά κυρίως την απαλλαγή του 2010, όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος δηλαδή. Γι' αυτό θα ήθελα εδώ να αποφελθώ από αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε και να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας και Δικαιωμάτων Καταναλωτών για την στήριξή σας σε αυτό το θέμα. Αυτή η αξιολόγηση είναι κάτι αναγκαίο για την ανεξαρτησία μας, διότι η ΕΦΣΑ έχει, όπως λέει η έκθεση, ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό βέβαια. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν ε, εφησυχάζουμε γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη στη δουλειά μας. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την νέα μας πολιτική και τους εφαρμοστικούς κανόνες που άρχισαν να ισχύουν τον Ιούλιο και να σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματά μας με μεγαλύτερη ακόμα σαφήνεια. Οι δράσεις μας επίσης καθοδηγούνται από τις συστάσεις της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου για την ανεξαρτησία κάποιων ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως επίσης και από τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Η ΕΦΣΑ, πολύ σωστά, είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της. Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα περισσότερη δουλειά μένει να κάνουμε και ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε είναι δύσκολο και σκληρό. Όπως πολύ σωστά εντοπίζει η έκθεση, η δουλειά μας είναι όλο και περισσότερη και μέσα σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον. Υπάρχει νέα τεχνολογία, υπάρχουν τα επιστημονικά επιτεύγματα και δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο όριο στις δυνατότητές μας να δώσουμε αξιολόγηση κινδύνου. Για παράδειγμα, η συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα για τις επιπτώσεις που έχουν μικρές δόσεις παραγόντων ή ενδοκρινικοί παράγοντες ή χημικά μείγματα. Τελευταία δημοσιεύθηκε κάτι για την ε, τοξικότητα των παρασιτοκτόνων και για παρασιτοκτόνα που δεν μπορούν να προστεύσουν μη γενετικά, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμεθα είναι επίσης όλο και πιο δύσκολο. Ο... οικονομική συγκυρία επίσης δημιουργεί βεβαιότητα. Επιπλέον, ελέγχεται το έργο μας όλο και περισσότερο προκειμένου να είμαστε πραγματικά αμερόληπτοι. Σαν ένας ε, δημόσιος οργανισμός που είμαστε, για μα ο έλεγχος αυτός είναι πρόσδεκτος. Οι συστάσεις στην έκθεση πάντως μας βοηθούν να επιβεβαιώσουμε τις μελλοντικέ μας προτεραιότητες, τις οποίες και θέλω να συζητήσω μαζί σας εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον ανοιχτό χαρακτήρα του οργανισμού μας και τη διαφάνεια και να βασιστούμε σε συναντήσεις ανοιχτές σε παρατηρητές και τα δεδομένα μας επίσης να κυκλοφορούν ευρύτερα. Είναι σαφές ότι η έκθεση τονίζει πως η ΕΦΣΑ μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα στη διεθνή σκηνή και να κάνει την ευρωπαϊκή φωνή να ακουστεί ακόμα περισσότερο σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Ενώ λοιπόν εμείς προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσεις όπως ήταν εκείνη του e-call στη Γερμανία και στη Γαλλία το 2011, συγχρόνως προσπαθούμε να εντοπίσουμε και αναδυόμενους κινδύνους πριν αποτελέσουν πραγματικό κίνδυνο για τις κοινωνίες μας. Η επιστημονική συνεργασία επίσης είναι ιδιαίτερα θετική και αποτελεσματική, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε το βήμα μας. Ερευνούμε και προσπαθούμε να έχουμε προπολογισμό για να κάνουμε και προπαρασκευαστική δουλειά και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία από εθνικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να βελτιωθεί και η ικανότητα αξιολόγηση κινδύνου μέσα στα κράτη-μέλη. Τώρα πρέπει να δούμε πώ θα εισάγουμε νέα μεθοδολογία και νέα εργαλεία, όπω είναι προγράμματα κατάρτιση και ανταλλαγέ πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να ισχυθεί η ιδέα τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα αξιολόγηση Κινδύνου. Η εξολόγηση επίσης συστήνει να αυξήσουμε την χρησιμότητα των επιστημονικών μας αποτελεσμάτων και θέλουμε όντως να τα κοινοποιήσουμε ευρύτερα, ώστε να ληφθούν κατάλληλε αποφάσεις. Κάποια από τα έγγραφα με κατευθύνες γραμμές που ετοιμάζουμε εμείς θα μπορούσαν να έχουν πιο εύχρηστη μορφή για τους χρήστες. Επιπλέον θέλουμε να ε, ανακοινώνουμε επιστημονικές συμβουλές με έναν πιο σαφή και απλό τρόπο. Γι' αυτό και πρόσφατα ε, οργανώνουμε την, ε, ξεκινήσαμε την οργάνωση της ΕΦΣΑ έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή. Όλα αυτά βέβαια δεν φτάνουν από μόνα τους, γιατί τα δικά μας πάνελ μπορεί να δίνουν αποτελέσματα, αλλά πολλοί εμπειρογνώμονες έχουν ιδιαίτερα φόρτο μεγάλο εργασίας. Εμείς αγωνιζόμαστε δηλαδή με διάφορα αριθμιστικά πλαίσια και μέσα σε αυτά πρέπει να ενισχύσουμε τους εμπειρογνώμονες γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τον κίνδυνο. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ικανότητας της ΕΦΣΑ. Έχουν γίνει κλήσεις και από το Κοινοβούλιο να κάνουμε ακριβώς αυτό, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα και των κρατών μελών για την αξιολόγηση κινδύνου. Αυτό θέλουμε να το λάβουμε υπόψη μας για το 2013 και μετά, αλλά χρειαζόμαστε τη δικιά σας στήριξη γι' αυτό. Μετά από 10 χρόνια εμπειρία της ΕΦΣΑ, θα ήταν σωστό να πούμε ότι η επιστήμη πολύ σωστά αποτελεί ένα ζωτική σημασία σε στοιχείο για την ε, πολιτική ασφάλεια τροφίμων. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτή που έχουμε στους ε, ώμους μας και την έχουμε αναλάβει ευχαρίστω. Ξέρουμε ότι συνεργαζόμενοι μαζί σας και με τους υπόλοιπους εταίρους μας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των εργασιών της ΕΦΣΑ. Συγχαρητήρια και για την δεκαετή, τα, τα γενέθλιά σας δεκαετία σας το πω έτσι, τα δέκα σας χρόνια που θα γιορτάσετε σύντομα και θα δώσω το λόγο τώρα στις και στους συναδέλφους μου για τοποθετήσεις και ενδεχομένως ερωτήσεις. Ο κύριος Πλίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εκτελεστική διευθύντρια της ΕΦΣΑ για την παρουσίαση του έργου του, του οργανισμού της θα υπογραμμίσω και αυτά που είπε ο πρόεδρος μας κύριος Γκρότε, ότι το έργο της είναι σημαντικό και ότι συντρέχει τις χώρες σε περίπτωση κρίσεων, όπως τώρα στην περίοδο αυτή της κρίσεως. Και βέβαια και στην ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία που προ δύο ετών είχαμε εκείνη την ε, έντονη κρίση όπου ε, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές από εκείνο το ε, μικροοργανισμό που βρέθηκε σε σαλάτες και η δράση της ΕΦΣΕ ήταν σημαντική. Συζητήθηκε πολύ στον τύπο εάν θα ερχόταν η κυρία Φρούβεν στο εκτελεστικό όργανο της ΕΦΣΑ. Το Κοινοβούλιο αντέδρασε και το απέτρεψε αυτό. Μετά βέβαια έπαυσαν οι δημοσιογραφικές φωνές όταν το σκάνδαλο λύθηκε και έπαυσε να υπάρχει. Έχουμε μερικές, μερικά εργοτάξια, στο πω έτσι, τα οποία ίσως θέτουν σε κίνδυνο το κύρος της ΕΦΣΑ στα μάτια του κοινού, αλλά δεν φταίτε εσείς. Όταν η προεδρεύουσα του Συμβουλίου μετακινείται σε άλλο οργανισμό, τότε που είναι άσχετος, τότε εμείς πρέπει να ασκήσουμε τη σχετική πίεση και, και το κάναμε. Η συγκεκριμένη μου αίτηση, το συγκεκριμένο αίτημα, είναι να εγκύψετε περισσότερο στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πολλά θέματα που είναι αρμοδιότητα της ΕΦΣΑ έχουμε την εντύπωση ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θεωρούν ότι α, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Δεν έχουν ομάδες πίεσης όπως Φεραίρο ή Νεστλέ. Γι' αυτό στις μικρές και, και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να εξηγήσετε τι συμβαίνει. Και γι' αυτό άλλωστε είχαμε ζητήσει στο εκτελεστικό σας συμβούλιο να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Και ένα δεύτερο θέμα, μια ερώτηση δηλαδή για το θέμα των ε, διατροφικών προφίλ. Έμαθα ότι η ΕΦΣΑ αρνήθηκε να τα εγκρίνει διότι και οι ίδιοι επιστήμονες δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιο ποσοστό περιεκτικότητας λιπαρών ή ζάχαρης και ούτω καθεξής είναι υπερβολικό. Σας παρακαλώ να το επιβεβαιώσετε ή να το απορρίψετε. Είναι αλήθεια ότι η ΕΦΣΑ είπε ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για αυτά τα διατροφικά προφίλ ή εσφάλουν οι πληροφορίες μου. Καλά, θα ακούσουμε και τις άλλες ερωτήσεις και έχουμε και ένα τηλεοπτικό team εδώ που έχει προσκαλέσει η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Λεπάζ. Νομίζω ότι, το, ότι η τηλεοπτική ομάδα λήψεων είναι η France 3, η οποία κάνει λήψη εικόνων. Επίσης από το Nouvel Observateur. Η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Διευθύντρια που ήρθε σήμερα να μας μιλήσει και να μας παρουσιάσει και το πώς έχουν τα πράγματα και τους στόχους του οργανισμού σας. Ανοιχτό πνεύμα, διαφάνεια. Νομίζω ότι η κατεύθυνση που ακολουθείτε είναι πραγματικά πολύ σωστή. Ελπίζω και εσείς να είστε ικανοποιημένοι από την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και με σημειώνει και ο Ernst Jung ε, σε έκθεσή του, η οποία μας απεστάλλει πριν από λίγους μήνες. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις, κύριε Διευθύντρια. Δεν θα εκπλαγείτε. Με αφορμή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε χθε. Μελέτη. Έναν γενετικό στροποποιημένο οργανισμό, τον ΝΙΚΑΠΑ 603, και που ε, εντοπίστηκε σε ένα φυτοφάρμακο. Είμαστε αρκετοί όσοι αναρωτιόμαστε γιατί ενώ η οδηγια 2018 απαιτεί την ανάλυση των ε, μακροχρόνιων επιπτώσεων ε, των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην ανθρώπινη υγεία, μέχρι τώρα δεν έχει απαιτηθεί και δεν έχει διαταχθεί καμία μελέτη. Ούτε έγινε βέβαιος από την πλευρά των όσων ε, εμπορεύονται του γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Έπειτα, μας είπατε ότι θα γίνουν και, αντι... και από την άλλη πλευρά ε, εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες εμπειρογνωμοσύνης. Όμως, εφόσον αυτός ο αραβόσιτος επετράπει να καλλιεργείται, δεν μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους επίσης να ζητούμε να αξιολογήσουν τη δουλειά τους. Είναι αντίφαση. Για λόγους λοιπόν δεοντολογικούς, τους οποίους και εσείς αναφέρατε, και με πνεύμα μεταρρυθμιστικό όπως και εσείς ε, έχετε υποσχεθεί εδώ και κάποιους μήνες, ότι θα προχωρήσετε προ αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω να θεσπίσετε ένα πάνελ, μια ομάδα ειδικών, τελείως ανεξάρτητο από εκείνου που έκαναν την πρώτη εκτίμηση και αξιολόγηση. Και θέλω να ολοκληρώσω λέγοντα ότι περισσότερο από ποτέ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειαζόμαστε έναν οργανισμό με πολύ ισχυρέ ειδικέ γνώσει. Τα θέματα τη δημόσια υγεία ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο και έχουν και οικονομική διάσταση πολύ περισσότερο από ποτέ πριν. Όλοι οι Ευρωπαίοι στι οικογένειε του αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ο καρκίνος ή οι εκφυλιστικές ασθένειες. Εδώ πολλαπλασιάζονται οι παθήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολίτες και πραγματικά υπολογίζουμε στον οργανισμό για να μας βοηθήσει όλους συλλογικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες υγείας και διαβίωσης των πολιτών μας. ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ κύριε Λιλάν για την ε, προσέλευσή σας και εγώ. Έχω μια ερώτηση να σας θέσω. Γιατί για τα ενδοκρινικά στοιχεία ως συστατικά Υπάρχουν, και το γνωρίζουμε, βιολογικές συνέπειες. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε κάποια τροποποιημένα γενετικώς προϊόντα. Άρα θα εξακολουθήσω στην ίδια οδό με τις προηγούμενες ερωτήσεις. και ήθελα εδώ να αναφερθώ και στην ε, διατροφική, τα διατροφικά χαρακτηριστικά είναι και αυτά σημαντικά. Θα μπορούσαμε να προσδώσουμε συγκεκριμένες αξίες στις δοσολογίες, την σύνθεση των ε, τροφίμων, εάν θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη διατροφή ή στις εβδομαδιαίες συνιστόμενες δόσεις, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια ισορροπία διατροφική. Η ΕΦΣΑ θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μέρος του πεδίου αρμοδιοτήτων της και η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την ένδειξη της ημερομηνία λήξης, της προθεσμίας που αναγράφονται στα τρόφιμα δηλαδή. Εδώ χρειάζεται κάποια διαδικασία που να καλύπτει τόσο τον καταναλωτή, αλλά και να μπορεί να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων, κάτι που τώρα συμβαίνει. Η συσκευασία ή μάλλον ε, το σύνολο του προϊόντος κάποιες φορές ε, καταλήγει στα, στον κάδο απορριμμάτων στο τέλος της, στην καταληκτική ημερομηνία. Δεν θα μπορούσατε να εκπονήσετε κάποια μελέτη που να μας δώσει νέες ιδέες όχι να διακυβευτεί βεβαίω η επιστημιστική ασφάλεια, αλλά να έχουμε καλύτερη διαλογή. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Η κυρία Λιωτάρ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Χισλέν που ήρθε σήμερα εδώ. Πράγματι υπάρχει διαφορά με την ΕΦΣΑ τότε που ήμουν το σημείο επαφή με την ΕΦΣΑ. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και όσον αφορά την ανεξαρτησία επίσης ξέρουμε ότι αρχίζει και στέκεται στα πόδια της. Έχω δύο ερωτήσεις παρακαλώ για κάποια θέματα τα οποία επιστημονικά θα ερευνήσετε. Μιλήσατε για το MK, το παράγοντα αυτόν και είπατε ότι θα ερευνήσετε πολύ για το θέμα αυτό. Ρώτησε και η κυρία Λαπάς εξάλλου. Το ίδιο λοιπόν θέλω και εγώ να ρωτήσω. Υπάρχει και κάποιος άλλος παράγοντας για τον οποίο επίσης θα κάνετε νέα αξιολόγηση διότι έχουμε 270 μελέτες από τις περισσότερες από τις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την ε, υγεία και έχω ακούσει από επιστήμονες ότι και με ένα ελάχιστο ποσό δημιουργείται διαταραχή ορμονική. Τι θα κάνετε λοιπόν. Ξέρω βέβαια ότι οι έρευνες χρειάζονται χρόνο. Πρέπει να γίνει μια καλή έρευνα, άρα χρειάζεται πολύς χρόνος. Όμως και όλες αυτές τις έρευνες και για το NK603 και για την βυσφινόλη α μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο η άφησα κάποια στιγμή θα μπορέσει να δώσει κάποια διάγνωση έτσι ώστε όχι απλώς να ενημερωθεί η Επιτροπή αλλά να υπάρξει ενδεχομένω ένα μορατόριο. Είναι δυνατόν η ΕΦΣΑ να το κάνει κάτι τέτοιο και αν ε, μπορεί θα το κάνει ή όχι και γιατί. Και αν πείτε πως δεν θα το κάνουμε για αυτές τις ουσίες τότε θέλω να ρωτήσω υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο στην ΕΦΣΑ, κάποια συμφωνία που αν μη τι άλλο να μπορεί να στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Φλόρεντς. Δεν είμαι ειδικό για τέτοια θέματα, αλλά πάντως έμαθα ότι προ λίγων ετών, πριν αναλάβετε εσείς, έγιναν πραγματογνωμοσύνες από πραγματογνώμονες, πώς να το πω, υπονομεύονταν λόγω συμμετοχής τους σε κάποια βιομηχανία, κυρίως από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτά τώρα έχουν διευκρινιστεί από εσά και καλά κάνατε. Τι είχε κάνετε όμως με τις πραγματογνωμοσύνες και μελέτες που συντάχθηκαν τότε. Συνεχίζονται αυτές ακούω με μεν από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία ότι συνεχίζονται οι πραγματογνωμοσύνες αυτές, ότι ισχύουν δηλαδή και ότι η βιομηχανία αυτή δρά με βάση αυτές. Η βιομηχανία, είναι η ερώτηση μου, έχει τη δυνατότητα να σας υποβάλει ε, κάποια σχόλια γραπτός και να ζητήσει την άποψή σας. Δηλαδή, μου είπαν ότι σοβαρές βιομηχανίες δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας και να σας θέσουν ερωτήσεις. Μπορείτε ίσως να μου πείτε ότι δεν είναι έτσι, αλλά βέβαια μπορώ και, μπορούμε, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν είναι όλες ε, οι βιομηχανίες ε, ύποπτες κάποιων κακών προθέσεων. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους συγκεγραμμένους. Θα παρακαλέσω λοιπόν την κυρία Διευθύντρια να λάβει ξανά το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις που της ετέθηκαν. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα, ευχαριστώ τον κύριο Λίζε για τα όσα είπε για το σημαντικό έργο της ΕΦΣΑ και που αναφέρθηκε και σε την υποστήριξη που δόθηκε σε πλήρωνες χώρες μέλη και στη Γερμανία για τον, για τον μικροοργανισμό, για τον Ιόλ Νικολάη. Θα αναφερθήκατε επίσης στην παροχή υποστήριξη σε μικρές και μεσές επιχειρήσεις και είπατε ότι ενδεχομένως οι ανησυχίε τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως για παράδειγμα είπατε με συμμετοχή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ. Βεβαίως γνωρίζετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, ΕΦΣΑ, της καθορίζεται με τον ιδρυτικό κανονισμό της. Έχουμε ένα ιδιαίτερο Διοικητικό Συμβούλιο με την έννοια ότι δεν έχουμε εκπροσώπους χωρών μελών, έχουμε 15 μέλη που περιλαμβάνει ένα εκπρόσωπο της Κομισιόν και το κριτήριο για, την, ε, για τον διορισμό τους εκεί είναι η ιδιαίτερη πραγματογνωμοσύνη τους, η ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη τους μάλλον, στη, σε θέματα ασφάλειας διατροφής. Τώρα υπάρχουν και σύμβουλοι, αλλά ίσως εκεί μπορεί να ληφθεί υπόψη η ε, πρότασή σας. Σημαντικό επίσης είναι να λεχθεί ότι την προσοχή μας στρέφουμε και στη βιομηχανία με την έννοια ότι λαμβάνουμε πολλές αιτήσει. Θεωρούμε ότι τα δύο τρίτα των εκροών μας κατευθύνονται σε ρυθμιζόμενα προϊόντα. Αυτό δεν υπήρχε απαραίτητα από τις απαρχές της ΕΦΣΑ, αναπτύχθηκε σιγά σιγά και γι' αυτό είναι σημαντικό που η ΕΦΣΑ υποστηρίζει και τους καταναλωτές αλλά και την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Εμείς εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τον απαραίτητο διάλογο και διάδραση και επανέρχομαι στα όσα είπε ο Φλόρεντς όπου κατανοώ την ερώτηση και τη δήλωσή σας ότι εννοείται δηλαδή ότι η ΕΦΣΑ πρέπει να δίνει ανεξάρτητες επιστημονικές απόψει, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να διατηρεί ένα όριμο και ευφυή διάλογο με την βιομηχανία και ιδίω με όσου υποβάλλουν αιτήσει σε εμά. Πρέπει δηλαδή να συνεννοούμεθα μαζί του, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνουμε τα σωστά δεδομένα και θα μπορούμε βεβαίω να τα αποκρινόμαστε στα καθήκοντά μα. Βεβαίω αυτό το εξασφαλίζουμε και ιδίω με την μονάδα αιτήσεων που δημιουργήθηκε πέρσι, Application Desk Unit, για να φροντίσουμε να έχουμε επικοδομητικό, να διεξάγουμε δηλαδή επικοδομητικό διάλογο με την βιομηχανία, με ανταλλαγή δεδομένων και βεβαίως οι δικές μας επιστημονικές μελέτες παραμένουν ε, ανεξάρτητες. Για την κυρία Λεπάζ, αναφερθήκατε σε μια μελέτη, στην οποία αναφέρθηκα και εγώ στην εισαγωγική μου ομιλία, και πράγματι επιβεβαιώνω ότι θα εγκύψουμε στο θέμα. Ήθελα επίσης να πω εν προκειμένου ότι ναι μεν είχαμε ακόμη λίγο χρόνο για να μελετήσουμε το άρθρο, αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν πρόκειται μόνο για το NK603, αλλά και για άλλα και για αυτήν την υπόθεση θα χρειαστώ λίγο χρόνο βέβαια για να συνεργαστώ με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες και τους άλλους εμπειρογνώμονες. Νομίζω πάντως ότι θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με τους ε, ειδικού του πάνελ των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αλλά και των ζυζανιοκτώνων για να δούμε αν υπάρχουν αποτελέσματα ε, τα οποία μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο ενδοκρινικό σύστημα. Για να το πω πιο απλά, θα εξετάσουμε προσεκτικά τη μελέτη, θα δούμε ποιοι είναι οι τομείς αρμοδιότητας δικής μας που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε τη μελέτη. Θα προχωρήσουμε σε διάλογο με τους συντάκτες της μελέτης για να μας διαθέσουν και έναν αριθμό ας πούμε, ομών δεδομένων, ανεπεξέργαστων δεδομένων, ε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εγκύψουμε στο θέμα. Λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο πάνελ των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών να εργαστούν στο θέμα δηλαδή, διότι έχουν ήδη εργαστεί στο θέμα. Αυτό που τους ζητούμε εμείς εδώ είναι όχι να επαναξιολογήσουν τη γνωμοδότησή τους, αλλά μια νέα μελέτη που μου φαίνεται μάλιστα αρκετά περίπλοκη και που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα προσεκτικά. Δεν βαίνει λοιπόν αντίθετα με την βασική αρχή που έχουμε και που ορίζει ότι ο ειδικό δεν μπορεί να επαναξιολογήσει την εργασία του. Η ΕΦΣΑ οφείλει να εξετάζει τα θέματα και να μην αμφισβητεί τα ε, ε, αποτελέσματα στα οποία έχει ήδη καταλήξει. Τώρα, για την αξιολόγηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έχουν περιγραφεί καθαρά στο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών μας, Guidance Document. Αυτές οι Guidance αναθεωρούνται τακτικά και για τρόφιμα, ζωοτροφές και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τους GMO υπάρχει εξέταση ανά περίπτωση στη βάση των κριτηρίων αυτών και είναι δυνατόν να ζητήσουμε πρόσθετα δεδομένα καθώς και τις μελέτες για παράδειγμα διατροφής των ε, αρουραίων σε ένα μακρότερο χρονικό διάστημα από ε, αυτό που ήταν συνήθως παλαιότερα ή σε άλλες μελέτες. Τώρα για το εάν ε, η μελέτη θα γίνει για 180 ημέρες ή για ε, μακρύτερο χρονικό διάστημα ε, όπως δύο ετών θα πρέπει αυτό να εξεταστεί. Είδαμε και τη μελέτη που συζητήθηκε χθε και μάλιστα προ λίγων μηνών είχε, είχε δημοσιευτεί και άλλη μελέτη που συνέκρινε τα αποτελέσματα της μελέτης 180 ημερών με τις μελέτες, δηλαδή, με τις μελέτες των δύο ετών και ε, έκρινε ότι η μελέτη των 180 ημερών επέτρεπε να προβλεφθούν ορισμένα, ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Βέβαια εγώ δεν έχω προσέλθει εδώ για να ε, εκφράσω άποψη για τις μελέτες αυτές. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει με σοβαρότητα και εμείς θα εγκύψουμε σε αυτήν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Και βεβαίως, όπως είπα, θα έλθουμε σε επαφή με τους συντάκτες της μελέτης αυτής για να συζητήσουμε μαζί τους. Ευχαριστώ βεβαίως και για τα όσα είπατε για την αναγκαιότητα οι οργανισμοί που ασχολούνται με την υγεία να είναι ισχυροί και σε ένα πλαίσιο βεβαίως όπως είπατε και εσείς οικονομικής κρίση, ε, ε, κρίσης που βεβαίως δεν πρέπει να λησμονείται ότι εάν κανείς χαλαρώσει την προσοχή του πράγματι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες στο μέλλον σε ό,τι αφορά τη δυσφενόλη ε, ε, αναμένουμε την πλήρη ε, εξέταση και όπως είπατε κυρία Λιωτάρ μελετούμε κάποιες εκατοντάδες νέων επιστημονικών δημοσιεύσεων από την περίοδο 2006-2012, άρα είναι πολύ εκτεταμένο το έργο αυτό, γιατί τη δυσφενόλη Α αναμένουμε να μπορούμε να έχουμε άποψη τον Μάιο του 2013 για να μπορέσει να ληφθεί απόφαση. Σωστά είπατε, την βάλατε μάλλον, την ουσία αυτή σε ευρύτερο πλαίσιο των endocrine disruptors ή των ενδοκρινικών ενεργών ουσιών που είναι ουσίες που ορισμένοι επιστήμονες έχουν προωθήσει την υπόθεση, έχουν καταθέσει ας πούμε την υπόθεση ότι ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην υγεία μας ακόμα και όταν είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο ενώ μπορεί να μην έχουν αρνητική επίδραση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι κλασική δυτικά μπύλη για, που ισχύει για ορισμένα χημικά, ορισμένα χημικέ ουσίε. Τώρα εδώ πρέπει να πω ότι πρόκειται για σημαντική πρόκληση για τους επιστήμονες να εργαστούν δηλαδή επ' αυτού. Δεν είμαστε μοναδικοί που εργαζόμαστε επί του θέματος. Πολλές δραστηριότητες αναλαμβάνονται και από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και από άλλες συνεργαζόμαστε δε στενά με τα πρόσωπα αυτά, με την EA και MEA, καθώς και της Non-Food Committee της ΣΑΝΚΟ. Λάβαμε νέα εντολή πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, που μας ζητεί να μελετήσουμε τις ενδοκρινικές ενεργές ουσίες, βεβαίως σε σχέση με τα τρόφιμα και ζωοτροφές, γιατί εκεί εντοπίζεται η εντολή μας, και θα μπορέσουμε να δώσουμε, να καταθέσουμε τις μελέτες μας τον επόμενο Μάρτιο με δήλωση της Επιστημονικής μας Επιτροπής όπου θα καταγράφουμε την πρόοδο την επιστημονική, της επιστημονικής γνώσης στο θέμα αυτό και να καταστρώσουμε επιστημονικά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οριστούν αυτές οι ενδοκρινικές ενεργές ουσίες. Τα τοξικολογικά τεστ που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι επαρκή για να αποκαλύψουν ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις των ουσιών αυτών. Καθώς επίσης θα συζητήσουμε και οποιαδήποτε άλλη σχετική σύσταση. Λέω ότι είναι σημαντική πρόκληση, διότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, όχι μόνο στην, μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας, αλλά και μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας. Έτσι λοιπόν εμείς θα κάνουμε μια καταγραφή της επιστημονικής γνώσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ για τα ε, ζυζανιοκτώνα που έχετε εσείς εγκρίνει κανονισμό μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών και ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ε, μελέτη για τον ρόλο, τον ενδεχόμενο ρόλο των ζυζανιοκτώνων επί των ενδοκρινικών ενεργών ουσιών. Αυτός φαντάζομαι ότι είναι ο λόγος για τον οποίο μας ζητεί άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσουμε αυτές τις προθεσμίες. Νομίζω ότι απάντησα και στον κύριο Λόρενς και για τον κύριο Πρόντι, για τον κύριο Φλόρενς, η Γενική Διευθύντρια. Αν υπάρχει και τίποτε άλλο βεβαίω που επιθυμείτε να μάθετε ασφαλώς θα επανέλθω. Γιατί τη δυσφενόλη δεν απάντησα στην υπόθεσή σας για το μορατόριουμ. Για την ώρα από όσο γνωρίζουμε, θα δούμε βέβαια πού θα καταλήξει το έργο μας, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία να υπαγορεύουν την θέσπιση πλήρους απαγόρευσης ε, χρήσης της ουσίας αυτής. Παρόλο που δεν αποφεύγουμε να τέτοια σύσταση, βεβαίως την τελική ευθύνη θα την φέρουν οι risk manager που περιλαμβάνουν βεβαίως και εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Εδώ έληξε η συζήτηση. Εγώ δεν έχω άλλους εδώ εγγεγραμμένους. Οι συναδελφοί μου έθεσαν ερωτήσεις. Βλέπω παρόντες και ορισμένους γενικούς, ε, και ορισμένους ε, συγγνώμη, επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα μεταξύ του κοινού παρακολουθεί τη συζήτησή μας. Παρό, παρότι ήταν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίω αυτό δείχνει ότι η δουλειά δεν τελείωσε εδώ. Συνεχίζεται. Ε, γιορτάζει τα δέκα της χρόνια η ΕΦΣΑ φέτος. Της εύχομαι καλή επιτυχία. Και βέβαια για τα 18 σας χρόνια θα περάσει λίγος καιρός ακόμα. Θα σας παρακολουθούμε, θα παρακολουθούμε την εργασία σας, βέβαια με κριτικό πνεύμα, αλλά θετικό. Και βέβαια με τρόπο που να διασφαλίζει μια δίκαιη αντιμετώπιση των μεν από τους δε. Κάτι που ίσως δεν υπήρξε πάντοτε τους τελευταίους μήνες. Είπαμε ότι θα παρακολουθούμε το έργο σας με κριτικό πνεύμα, αλλά δίκαιο. Είμαστε υπερήφανοι για του οργανισμού μας και μια φορά λησμονούμε ότι είναι ανεξάρτητοι και κάτι που συζητείται συχνά ότι η επιστήμη και οι εμπειρογνώμονε πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, αυτό είναι πραγματικά μια επιταγή. Καμιά φορά βέβαια κινείται κανεί στην κόψη του μαχαιριού, διότι θέλουμε να έχουμε και επιστήμονε οι οποίοι να είναι καλά δικτυωμένοι και να έχουμε στη θέση μα του καλύτερου επιστήμονες. Πρόκειται για μια προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου με κανόνα και διαβήτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς βεβαίως θα σταθούμε στο ύψος μας ως θετικοί αλλά αυστηροί κριτές του έργου του οργανισμού σας. Όπως είπατε και εσείς έχουμε ακόμη πολλή δουλειά και έχουμε βεβαίως τις νέες τεχνολογίες, νέες ουσίες, νέες παραγωγικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας. Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler ο επιστήμον που είναι προσκεκλημένος εδώ σήμερα θα ήθελε να συνεχίσει την συζήτηση με την κυρία Δεπάζ και με το τηλεοπτικό συνεργείο εκτός της αιθούσης. Διότι έχουμε και δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα με την Γενική Διευθύντρια κυρία Μακλέιντ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που καλωσορίζω σήμερα εδώ και δηλώνω την ικανοποίησή μου που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί της για την πρόοδο των εργασιών του οργανισμού της. Έχει το λόγο για να παρουσιάσει την εργασία του οργανισμού της. Σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να έρθω και να ανταλλάξουμε απόψεις για το έργο του οργανισμού και σα ευχαριστώ για τη στήριξη του Κοινοβουλίου και των κατών μελών. Νομίζω έχουμε ένα κοινό στόχο να έχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους πολίτες της Ευρώπης. Οι δύο οργανισμοί, ο οργανισμο για τα Τρόφιμα και για το Περιβάλλον, κάποιες φορές έχουν ακριβώς την ίδια δυσκολία να συνδυάσουν σε κοινό πεδίο διαφορετικές απόψεις, αλλά συνεργαζόμαστε, όπως για τις ενδοκρινικές ενεργές ουσίες. Και ελπίζω να πετύχουμε και κάτι στο άμεσο μέλλον. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω εδώ και τους δύο εκπροσώπους που συμμετέχουν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, τον ε, κύριο Σκούλο και τον κύριο Χένικε, και είναι και ένα βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ τη Επιτροπή σα και του οργανισμού μα. Πολύ σύντομα, του τελευταίου μήνε, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε το έργο των εισηγητών, ιδίω τη Επιτροπή σα, για θέματα όπω το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον, η αποδοτικά των πόρων, διαφορετικέ πτυχέ τη βιοπικιλότητα, ε, η φύση και, τα, χημικέ ουσίε. Υπάρχει επίση μια κοινή πρωτοβουλία του Προέδρου για συστηματικό διάλογο μεταξύ των εισηγητών και των προσώπων των διαφόρων ενδιαφερομένων οργανισμών. Να ευχαριστήσω την, ε, τα μέλη της Επιτροπής για την ε, διαρκή στήριξη σε μένα προσωπικά αλλά και σε όλα τα μέλη του οργανισμού και στη διαδικασία της απαλλαγής για τον ε, περσινό προπολογισμό. Σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Όπως θα γνωρίζετε, ο οργανισμός ε, είναι στη φάση της πενταετούς ε, αξιολόγησής του, την οποία έχει αναλάβει η ΚΑΟΗ με, τα, με τις συμβάσεις πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και θα λάβει την τελική έκθεση κάποια στιγμή το 2013, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως προς τη στήριξη προς άλλες επιτροπές, ε, προσφέρουμε στήριξη και στην Επιτροπή Μεταφορών και Γεωργίας, και βεβαίως στοιχεία και υλικό για τις επισκέψεις των βουλευτών ε, σε διάφορες περιοχές όπως την Κύπρο. Στήριξη προσφέρουμε και σε άλλα μέλη άλλων επιτροπών και σε εθνικές συναντήσεις και συνέδρια όπως στο Ντέρμπαν και στο Ρίο Συνήκωση. Εκεί νομίζω ότι με άλλους οργανισμούς ε, είδαμε ότι έχουμε κοινούς στόχους και ότι το έργο που επιτελέσαμε στην Ευρώπη το έργο που, που, επιτελέσαμε στην Ευρώπη και ονομάζεται το βλέμμα στραμμένο στη γη είναι κάτι που έχει αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλου. Εδώ προσπαθήσαμε να ε, μοιραζόμαστε ζωτικέ πληροφορίε και αυτό είναι ένα τέταρτο πυλώνα τη δημοκρατία. Δεν είναι κάτι που το βάλουμε στο σιρτάρι οι πληροφορίε και τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε, αλλά πρέπει να το αξιοποιούν οι νομοθέτε ώστε να μπορούν να λάβουν τι σωστέ και τεκμηρωμένε αποφάσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η διεθνή προοπτική που έχουμε μπορεί να μα κάνει περήφανου. Και πολλέ από πολλοί από τους διεθνείς οργανισμούς και τα κρατη και οι φορείς βλέπουν ότι βρισκόμαστε στην πρωτοπορία. Παρομοίως, έχει αναγνωριστεί ότι και το έργο μας το πρόγραμμα GMES αλλά και η στήριξή μας στο GIO και το GEOSS ε, είναι πολύτιμο. Αυτό φάνηκε και στο Τζέτζου ε, όταν συναντηθήκαμε για την κατάρτιση του χάρτη για τις ε, χερσαίες υπηρεσίες. Και είδαμε πόσο σημαντική ήταν η δική μας συμβολή. Πάντως, για το πρόγραμμα GMES ε, χαίρομαι που ακόμη συνεχίζεται, ακόμη και αν θα επηρεαστεί από τη συζήτηση για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές, διότι τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν πλέον ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πολλά από αυτά που γίνονται και με τη διαδικασία τακτική υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση. Αυτά θα έχουν ε, επιρροή και στι ε, επενδύσει που θα γίνουν στο διάστημα και για το πώ θα καλύψουμε την ευρωπαϊκή επικράτεια και συνολικά τις χερσαίες υπηρεσίες παγκοσμίω. Εδώ θα φροντίσουμε και την συνιστόσα του GMS in situ, γιατί είναι πολύ σημαντική και η διάσταση των γεωδιαστημικών στοιχείων αναφοράς 24-7. Εδώ λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία που σε εθνικό επίπεδο δεν διατίθεται. Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον για το πρόγραμμα εργασιών του 2013. Να επαναλάβω ότι πραγματικά σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στις συζητήσεις περί προπολογισμού. Μα ανατίθενται ολένα και περισσότερε αρμοδιότητε μέσω τη νομοθεσία, με διάλογο με τα κάτι μελη με τι υπηρεσίε τη Επιτροπή. Χρειάστηκαν περαιτέρω κονδύλια, ιδίω για το θέμα τη κλιματική αλλαγή και τι σχετικέ πολιτικέ για την ατμόσφαιρα. Οι βασικέ μα προτεραιότητε για το 2013 είναι οι εξή. Η θεματική τη ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε να υπάρξει σημαντική μεταρρύθμιση εδώ στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και η προσαρμογή. Εδώ περιμένουμε μείζονε εξελίξει στο ερχόμενο διάστημα. Η αποδοτικότητα των πορών, η πράσινη οικονομία, το οικοσύστημα, η ε, καταγραφή των φυσικών κεφαλαίων. Επίσης, πώς θα μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση με το πρόγραμμα ICT, και βεβαίως το πώς κάθε χώρα εκτός πια Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης του 27, θα μπορέσει να εξαπλωθεί και στα Βαλκάνια, στη Σκανδιναδία, ε, στον Αρκτικό κύκλο και ούτω καθεξής. Θα δούμε τώρα τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της φετινής χρονιάς, γιατί πραγματικά είχαμε κρίσιμους διαλόγους και ανταλλαγή απόψεων. Και το θέμα είναι αν έχουμε αρκετά κονδύλια για να στηρίζουμε το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να πω έτσι εξ αρχή είναι ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή μα την πολυτέλεια να μην φροντίζουμε το περιβάλλον. Για την ποιότητα τη ατμόσφαιρα. Ο οργανισμό μα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων για την ποιότητα τη ατμόσφαιρα. Του ερχόμενου μήνε θα παρουσιάσουμε τα πιο πρόσφατα πορίσματα και θα δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να πετύχουμε του στόχου του ΠΟΗ. Όμω Πέρσι ε, δημοσίευσαμε μια έκθεση που δείχνει ποιο είναι το κόστος της ε, ζημιάς στην υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Οι 10.000 μεγαλύτερες ρηπογόνες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη κοστίζουν 169 δις ευρώ ε, ετησίως και αυτό προέρχεται από 191 μόνον μονάδες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ο βιομηχανικός κλάδος αναγνώρισε ο ίδιος, εφόσον εκεί ανήκουν αυτές οι 199 ε, μονάδες, ότι κάποιες φορές είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση του στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο οργανισμό συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ω προ την οδηγία NEC, την EPRTR και την οδηγία ID. Και το θέμα είναι να αναθεωρήσουμε και την ε, στατική για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολλές αντιστάσεις από τις χώρες για τις περαιτέρω προποθέσει που θέλουμε να θέσουμε. Εδώ όμω σαφώ θα πρέπει να, είμαστε, να δείξουμε πυγμή και πρέπει πραγματικά να επιτελέσουμε ακόμη πολύ πρόοδο. Η σύμβαση LRTAP επίσης μας ε, έχει απασχολήσει και την έχουμε προωθήσει και βεβαίω συζητούμε και με τις γειτονές χώρες, την Ομοσπονδία της Ρωσίας, τις ΗΠΑ, Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, προκειμένου να βελτιώσουμε τα δεδομένα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας της ποιότητας καθημερινά. Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να ανταλλάξουμε στοιχεία μαζί τους και είναι το ίδιο για τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Επίση, είναι πολύ σημαντικό και για τους πολίτε το τι γίνεται εκεί που ζουν, όπω για το όζον, όπως το, στοιχείο όπως το όζον, οι ουσίες οξύδωσης η ποιότητα της ατμόσφαιρας, ε, το τι γίνεται στα αστικά κέντρα. Σε συνεργασία λοιπόν με τα κράτη-μέλη ξεκινήσαμε πιλωτική μελέτη σε συνεργασία με τους πολίτες, ε, με διάφορες πόλεις μάλλον στην ε, Ευρώπη, το Βερολίνο, το Μάλμο, το Δουβλίνο, τη Μαδρίτη, την Πράγα, το Πλογέστη, τη Βιέννη, προκειμένου να βελτιώσουμε την εφαρμογή τη νομοθεσία. Στι πιλωτικέ αυτέ μελέτε συνεργαζόμαστε με τι δημοτικέ αρχέ, προκειμένου να καταγράψουμε τι τοπικέ εκπομπέ αερίων, το πώ κατανέμονται οι διάφορε πηγέ ρήπανση, ε, του σταθμού παρακολούθηση, την διαχείριση και το τι γίνεται με την ενημέρωση του κοινού. Τελικά οι πολίτε εκεί βλέπουν την αξία των ευρωπαϊκών οργανισμών στην καθημερινότητά του. Ο θόρυβο είναι ένα άλλο σημαντικό τομέα που απασχολεί πολύ του πολίτε γιατί έχει σημαντικέ επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία και εδώ με την καινοτόμο χαρτογράφησή μα νομίζω χάρη στη στήριξη βεβαίω των τοπικών αρχών και όλο και περισσότερε ομάδε που ενδιαφέρονται στην για την παρακολούθηση του θορύβου, ιδίω λόγω των μεταφορικών μέσων ή τα αεροδρόμια και άλλα συγκεκριμένα σημεία όπου ο θορύβο είναι αυξημένο, εκεί ε, καταφέραμε να έχουμε μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται στα smartphones και βεβαίω είναι ένα μέσο ιδιαίτερα σύγχρονο για την παρακολούθηση του θορύβου και την εξέλιξή του. Ομάδε πολιτών, τοπικέ αρχέ μα αποστέλνουν πληροφορίε και δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη χαρτογράφησή μα. Είναι λοιπόν πολύ πιο επικαιροποιημένη η χαρτογράφηση και πολύ πιο ρεαλιστική για το τι συμβαίνει εκεί που ζουν οι άνθρωποι και οι πολίτε και για το τι συμβαίνει με νέε εγκαταστάσει, μονάδε και υποδομέ. Για την κλιματική αλλαγή, όπως πολλοί θα γνωρίζετε, εδώ ε, έχουμε ασχοληθεί σοβαρά και με τις κλιματικές ε, πολιτικές και με τις ενεργειακές πολιτικές. Ε, προτείνουμε μέτρα τα οποία είναι και περισσότερο εγκρίνονται, όπως λόγω χάρη την έκθεση καταγραφής των αερίων του θερμοκηπίου που υποβάλαμε στην UNFCCC και ασχολούμαστε και την καθημερινή εργασία του και λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών. Ασχολούμαστε με την διοξίδιο του άνθρακα ε, και το πόσο αυτό εκπέμπεται από αυτοκίνητα και φορτηγά, ε, με τα αυτοριούχα αέρια και την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την κατανομή των προσπαθειών. Κοιτάζουμε τι γίνεται με την αεροπλοεία, βεβαίως και για τις εκπομπές στην αυσιπλοεία. Το θέμα είναι πώ θα εξασφαλίσουμε επίση ε, υψηλή ποιότητα δεδομένα. Η απόφαση για την κατανομή των ευθυνών και τα βασικά έτη που έχουν οριστεί είναι σημαντικά προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερα δεδομένα τα κράτη-μέλη. Εδώ είδαμε ότι το 50% των δεδομένων που είχαμε ω τώρα ήταν ε, μειωμένη ποιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα για να καταγράψουμε τα στοιχεία εκτό του συστήματο ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε στη σωστή αυτή κατεύθυνση, γιατί είναι κρίσιμο για τι προσπάθειε εκπαιδευτία που καταβάλει η Ένωση και σε διεθνέ επίπεδο να επιτύχουμε αποτελέσματα. Η ποιότητα, και ξανά η ποιότητα και πάλι η ποιότητα είναι ο πρώτο μα στόχο. Υπάρχουν όμω και καλέ ειδήσει για τι εκπομπέ των αερίων του θερμοκηπίου από τα τελευταία νέα που έχουμε. Είδαμε ότι έφτασαν κατά 2,5% το 2011 παρόλο ε, που αυξήθηκε η κατανάλωση του άνθρακα και αυξήθηκε και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Μάλιστα, εκεί που υπήρχαν κοινέ δεσμεύσει υπό το πρωτόκολλο του Κιώτο, ε, έπεσε κατά 3,5% το συνολικό ποσοστό εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Βλέπουμε ότι οι δεσμεύσει του Κιώτο βεβαίω δεν έχουν ακόμα πληρωθεί, όμω ήταν και ποιότερο ο χειμώνα και υπήρχε λιγότερη ζήτηση για ε, θέρμανση των νοικοκυριών και μικρότερη κατανάλωση φυσικού αερίου. Ήταν οι λόγοι που έπεσαν τα ποσοστά αυτά. Τώρα για τις για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα γεωταχή. Εδώ βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν όλο και περισσότερο αυτοκίνητα που είναι ενεργειακώ αποδοτικά και οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στα αυτοκίνητα καθημερινά πέφτουν ε, στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε όμως ακόμα περισσότερο να επιτύχουμε τους στόχους της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα τα, οι εκπομπές από τα αυτοκίνητα τα 135,7 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, ενώ το 2010 ήταν στο 4,6% διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, δηλαδή είχαμε μια μείωση μόνο του 3,3%. μια συνολική ανάλυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στον τομέα των μεταφορών είναι κάτι που θα το συμπεριλάβουμε στην έκθεση τέρμα το φθινόπωρο της φετινής χρονιάς. Ω προ την προσαρμογή στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη, έχουμε πραγματικά μια ψηφιακή πλατφόρμα ιδιαίτερα καινοτόμα, η οποία έχει αποτελέσει πηγή γνώσεων για το πώ ανταποκρίνονται οι χώρε στι υποχρεώσει του και πού βρίσκονται οι ελλείψει, οι ανεπάρκειε, τα επιτυχή αποτελέσματα. Βλέπουμε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση και διαχείριση των στοιχείων αυτών. Όλοι χρειάζονται πληροφορίε για τι κλιματικέ αλλαγέ και το πρέπει να κάνουν η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τι πλημμύρε λόγω χάρη, τι πυρκαγιέ είναι εξίσου σημαντικά και έχει μεγάλη ζήτηση. Ω προ τη βιοπικιλότητα, όπω θα γνωρίζετε, είμαστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση τη οδηγία για τα οικοσυστήματα και το Natura 2000. Υπάρχει πρόγραμμα δράση σχετικά και αυτό που προσπαθούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι η μείωση για πρώτη φορά τη ζημιά στα οικοσυστήματα τη Ευρώπη και του φυσικού τη κεφαλαίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Προσπαθούμε να, να καταρτήσουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία για αυτά ε, και με τα, με τα συστήματα καταγραφή οικονομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα του ΟΗΕ και βεβαίω σε συνεργασία και με την ε, Στατιστική Επιτροπή του ΟΗΕ πρέπει να δούμε τι γίνεται με του φυσικού πόρου ε, στου οποίου βασίζεται η οικονομία μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε μια σαφή εικόνα. Επίσης, μαζί με συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβλέπουμε την ανάγκη να υπάρξει στήριξη του έργου μας και στην ευρύτερη γειτονία της Ευρώπης. Όχι μόνο για τη βιοπικιλότητα και τους φυσικούς πόρους, όπου υπάρχουν μεγάλες, τεράστιες δυνατότητες και δυναμικό στη γειτονία μας, αλλά είναι καλό ότι διαπιστώνουμε καλή κατάσταση τη βιοπικιλότητα σε πολλέ περιοχέ. Αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτή τη αρχή, λοιπόν για τα συστήματα πληροφοριών, μέσω της υποβολή εκθέσεων, μέσω της χαρτογράφηση, του χαρακτηρισμού και της συμμετοχή των πολιτών. Για το νερό, καθοριστικό σημείο και θέμα για φέτος ε, και ε, με επιλογή τη Προεδρία. Θα συζητήσαμε με το αποτύπωμα και την θαλάσσια στρατηγική διάφορα κριτήρια για τα οικολογικά ε, δεδομένα, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή από τους ενδιαφερομένους. Και κάτι που έχει να κάνει και με την προηγούμενη συζήτηση. Τι θα γίνει με τι ενδοκρινικέ ενεργέ ουσίε και άλλα στοιχεία φαρμακευτικά, τα οποία μπορεί να φτάνουν και στο πόσιμο νερό ή στα συστήματα υδροδότηση. Τι γίνεται με τα συστήματα διήλυση. Και τι συστήματα επεξεργασία νερού έχουμε και πόσο αποδοτικά είναι. Αυτό που αναζητούμε πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι το κόστο. Το κόστο που βαρύνει τι υποδομέ και τι εγκαταστάσει τι πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, οι εταιρείε υδροδότηση και πώς θέλουμε να διαγραφεί το μέλλον. Ε, θέλουμε μια ποιότερη προσέγγιση ή περισσότερη μηχανική προσέγγιση. Ω προς το νερό επίσης έχουμε ευθύνε και για τα νερά όπου επιτρέπεται το κόλυμπι, αφού είναι μέρος τη ψυχαγωγίας ε, για τους πολίτες. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερω οι άνθρωποι για το θέμα αυτό και νομίζω ότι έχουμε πραγματικά αρκετά καλέ θάλασσε. Υπάρχουν πάντω και ανεπάρκειε. Αυτό πολλέ φορέ οφείλεται και στι πλημμύρε ή σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα για την αποδοτικότητα των πόρων, τι πρώτε ύλε, την ενέργεια, τα απορρίμματα, την παραγωγή και την καταλάρωση. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά για το θέμα αυτό, ιδίω με την παραγωγή δικτών για να καταγράψουμε συγκεκριμένε τάσει που διαμορφώνονται. Αλλά ένα από τα εμβληματικά βήματα που κάναμε είναι η ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος ως προς την αυξανόμενη ζήτηση για πρώτες ύλες και τους πόρους που χρειαζόμαστε από τις αναλύσεις μας. Είδαμε ότι η και η παραγωγή πρέπει να μα ευαισθητοποιήσουν ω προ την διαθεσιμότητα των πόρων και τι ίδιε τι πρώτε ύλε. Η έκθεση περιδικτών νομίζω ότι το υπογραμμίζει αυτό και πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των πόρων. Δεν είναι αυτή η μόνη απάντηση. Πρέπει να σκεφτούμε την αθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και από άλλε προοπτικέ. Και οι συσχετισμοί εδώ είναι πολύ σημαντικοί όταν θέλουμε να, θέσουμε, να καταγράψουμε συγκεκριμένα προγράμματα και στόχους. Επίσης, τονίσαμε την πίεση που θα βαρύνει την Ευρώπη, ιδίω ό,τι αφορά την κατανάλωση, τη χρήση διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και υλικών, ακόμη και αν πρόκειται για τις σπάνιες γέες ή το πόσο χρησιμοποιούμε τους πόρους μας. Φαίνεται ότι το κόστος των... τη υποβάθμιση των περιβαλλοντικών πόρων για την κοινωνία δεν έχει αποτιμηθεί σωστά ω τώρα και ω προ την τιμή των ε, εμπορεμάτων, των αγαθών και υπηρεσιών. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα χάσμα σε σχέση με την πραγματικότητα, όπω την ε, καταγράφουμε και το πώ ε, το αντιλαμβάνεται το κοινό. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη συζήτηση μαζί του, γιατί υπάρχουν και οικονομικέ πιέσει. Δεν μπορούμε να περνάμε μόνο σε, σε φορολογικά μέτρα αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί. Όμω η αποδοτικότητα δεν θα είναι η μόνη λύση. Θα πρέπει να επιδιώξουμε και δημοσιονομική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να βελτιώσουμε Τη προσπάθειε ανακύκλωση, να δούμε από πού προέρχονται τα υλικά που χρησιμοποιούμε, οι πρώτε ύλε και η πόρη μα, εάν θα αλλάξει η δημοσιονομική μα δομή ή θα αλλάξουν οι τάσει καταναλωτικέ. Έχουμε εκθέσει ε, και για αυτά τα θέματα. Γίνονται συζητήσει με πολλά κατημέλη για το πώ θα πρέπει να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση αυτή, για τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση και τα επιπλέον στοιχεία που θέλουμε να καλύπτει. Και είναι σαφέ ότι πολύ περισσότερα μπορεί να γίνουν για τα απορρίμματα. Έχουμε ασχοληθεί με τι αναλύσει εξ για την επεξεργασία των απορριμμάτων από τι διάφορε χώρε. Δεν είμαι βέβαιο ότι θα πετύχουμε, του στόχου πετύχουμε του 2020, βεβαίω. Όμω η υλοποίηση της, ε, των κανόνων για την επεξεργασία των απορριμμάτων και τη βιομηχανία ανακύκλωση είναι κάτι που θα μα απασχολήσει σαφώ. Κλείνοντα, ήθελα να πω ότι είτε μιλάμε για την ε, μεταφορά απορριμμάτων διασυνοριακά, νόμιμη ή όχι, ή μιλάμε για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει συνθετική επεξεργασία με παραγωγή όμως πολλών χημικών συστατικών που μπορεί να βλάπτουν το περιβάλλον, σε κάθε περίπτωση έχουμε κάποιες από τις πιο αμφιλεγόμενες εκθέσεις μας που αφορούν το θέμα αυτό. Η πιο γνωστή είναι εκείνη για τις ενδοκρινικές ενεργές ουσίες που συζητήθηκε πριν από δύο μήνες. Είναι μια ιστορία, ένα θέμα που είναι αρκετά θλιβερό γιατί βλέπουμε ποιες είναι οι επιρροές στο περιβάλλον, τι ζημιές προκαλούνται, ότι τα ζώα, τα φυτά, τα αμφίβια, τα ψάρια είναι εκτεθειμένα σε αυτούς τους προγόνε ουσίες και πολύ περισσότερα ακόμη μπορούν να γίνουν. Ακούσαμε την πρόσκληση τη ΕΦΣΑ να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν στενότερα μαζί του και να δίνουμε τι προσπάθειέ μα και έχουμε δίκιο. Το Δεκέμβριο η έκθεση που θα δημοσιεύσουμε, η τελική έκθεση που θα δημοσιεύσουμε και θα μα στηρίξετε σε αυτό, είναι το τι θα γίνει με συγκεκριμένε ουσίε όπω ο μόλιβδο, ο υδράργυρο, ε, ε, και για την έγκαιρη προειδοποίηση σε σχέση με αυτές τις χημικές ουσίες στο περιβάλλον μας. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει ακόμη να έχουμε κατά νου ότι πολλές φορές πληρώνουμε την αμελιά μας με, τη, με στην ανθρωπινή υγεία και στο περιβάλλον. Η έκθεση αυτή που μπορεί να φτάσει και τις 130 σελίδες αντιμετωπίζει, μάλλον καλύπτει συγκεκριμένα και μία προς μία όλες τις ε, ευθύνε που έχουμε και τους συγκεκριμένους κινδύνους τι γίνεται με ένα ανθρώπινο σώμα όταν ε, μέσα σε έναν ολόκληρο κύκλο ζωής μπορεί να έχει απορροφήσει τέτοιες ουσίες. Δεν έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένα νομοθετήματα που θα πρέπει να καλύπτουν το κάθε θέμα, όμως κοιτάζουμε πώς ευφυώς θα πρέπει να προβλέπουμε για τις επόμενους νομοθετικούς μας στόχους. Um- Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την εκτεταμένη παρουσίαση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Είναι βεβαίω ευρύ το πεδίο των θεμάτων που καλύπτεται και γνωρίζουμε επίσης ότι έχετε μεγάλη σεωρευμένη γνώση. Με ενδιαφέρει ε, η Επιτροπή μας και η οι συγητές μας να έχουν πρόσβαση στις γνώσεις αυτές, γιατί αυτό δεν είναι πάντοτε γνωστό. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι πάντοτε γνωστή στους εισηγητές. Πρόκειται λοιπόν για μεγάλες και σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ποικιλία θεμάτων. Μιλήσαμε και με την αποδοτικότητα χρήσεως των πόρων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν θα έχουμε και τους σχετικούς δείκτες, έναν υπέρτερο δείκτη, τους επιμέρους δείκτες και στο ενδιάμεσο πρέπει να είναι ε, τα οικονομικά κυκλώματα. Μιλήσαμε επίσης και για την COP18 χθες. Μου άρεσε επίσης το ότι κάνετε και εκ των υστέρων επεξεργασία των θεμάτων εξηγήσαμε πρόσφατα σε μια παρουσίαση ότι πρόκειται για το λεγόμενο reality check που δεν κάνει πάντοτε το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ που στο μέλλον πρόκειται να κάνετε και μελέτη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου. Διότι εμείς έχουμε υπολογίσει ότι κάθε χρόνο μπορούν να προστίθενται 400.000 νέες θέσεις απασχόλησης εάν ε, μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τις δηλώσεις σας. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους του Management Board. Ο κ. Κόλας είναι εδώ και ο κ. Χένεση. Ποιος θέλει πρώτος, αφού είστε εδώ, να σας δώσουμε την ευκαιρία να μας απευθύνετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μας ε, προσκαλέσατε και που μας δίνατε το λόγο. Η παρουσία μας πρώτα απ' όλα στο Management Board και οι συζητήσεις που γίνονται για την διατύπωση του προγράμματος εργασίας είναι μια μεγάλη ευθύνη. Μερικές φορές μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε, αλλά έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά από εσά και από τους προκατόχους σας ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι χρήσιμο για τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει συγχρόνως να είναι χρήσιμο και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για ολόκληρη την Ευρώπη και για την Ευρώπη ως κομμάτι που παίζει ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο οργανισμός μας λοιπόν προσπαθεί να συνεισφέρει στην διατήρηση της ισορροπίας αυτής και με αυτό το πρόγραμμα. Σε ένα μεγάλο βαθμό η φωνή της Ευρώπης σε διεθνή φόρα έτσι ενισχύεται, στηρίζεται από το έργο του οργανισμού. Στο πρόγραμμα αυτό βλέπουμε ότι θα συμβεί ακριβώς το ίδιο. Από την άλλη, υπογραμμίζεται όλος ιδιαίτερο η οικοδόμηση ικανοτήτων σε ορισμένους τομείς που χρειάζονται κάποιες χώρες. Και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με τη δουλειά του οργανισμού με τα εθνικά κοινοβούλια που δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, αλλά πάντως σε νέους ιδιαίτερα τομείς όπως είναι οι οικολογικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπως αυτή, για μερικές χώρες λοιπόν είναι η καλύτερη στιγμή προκειμένου να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στην οικονομία και την πράσινη οικονομία και τους φυσικούς πόρους τους οποίους πρέπει να βασίζεται η οικονομία αυτή. Γραπτά μάλιστα σας έχουμε στείλει και κάποια σχόλια. Προσπαθούμε συγχρόνως να δούμε σε πλανητικό επίπεδο την πράσινη οικονομία και σε αυτά τα πλαίσια πώς θα έχει ηγετικό ρόλο η Ευρώπη, διατυπώνοντας αν μη τι άλλο μία συνεκτική άποψη. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος και οι δικές μας εργασίες, αλλά και οι απαιτήσει. Δεν υπάρχει μόνο η οδηγία για τα ύδατα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ύδατα διασυνοριακά όπου υπάρχουν αλλαγές, ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα όπως είναι οι πλημμύρες. Και εκεί ακριβώς το πρόγραμμα πιστεύουμε του οργανισμού πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο. Θα ήθελα να δω λίγο και το θέμα του εδάφους. Θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, πιστεύω, στο πρόγραμμα αυτό. Ναι, δεν υπάρχει το θέμα της γης, αλλά νομίζω ότι θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί για την Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και θα ήθελα να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ο συνάδελφος νομίζω ότι μπορεί να συμπληρώσει αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σένινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Μάικλ. Είμαι νέος στο Management Board, αλλά από καιρό θαυμάζω το έργο που ασκεί ο οργανισμός, καθώς επίσης και η ηγεσία του. Εάν κανείς στρέψει τα βλέμματά του στον επιστημονικό κόσμο θα δει ότι ότι όντως μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τον οργανισμό αυτό και εμείς οι δύο αλλά και τα άλλα μέλη του Management Board παρακολουθούμε το έργο αυτό με κριτική, κριτικό υποστηρικτικό πνεύμα. Ο Μάικλ μίλησε για, το, για την επιστολή. Γιατί γράψαμε την επιστολή αυτή. Θα σας πω μαζί με μια παράκληση να δοθεί ίσως κάποια προτεραιότητα για την έρευνα, την, την έρευνα εφαρμογής, δηλαδή να παραχθούν μελέτες οι οποίες θα επιτρέψουν την επιτάχυνση των, ε, της έρευνας εφαρμογής. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία καθιστούν απαραίτητη την αντίδραση αυτή και να ενισχύσουμε την επιστημονική προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Το περιβάλλον και η επιστήμη βαδίζουν όλο και στενότερα, χέρι με χέρι. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε με ενοποιημένο, ενιοποιημένο τρόπο τους τομείς αυτούς. Όπως είπε και ο Μάικλ, δύο θέματα, η τρία, που αναφέρουμε στην επιστολή μας. Το Ρίο συν 20 κατέδειξε ένα πλήθος νέων ενιών, την green economy, green growth, inclusive growth, το decoupling και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε Έχουμε την ελπίδα ότι από τον οργανισμό θα μπορέσουν να γίνουν μεταέρευνες. Με την έννοια να εγκύψουμε να δούμε τι κάνει ο ΩΣΑ, τι κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα και τι κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Για να δούμε πώς θα περάσουμε από το περιγραφικό επίπεδο στο επίπεδο εφαρμογής. Παράγουμε δηλαδή δεδομένα, παράγουμε παράγοντες για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό το decoupling στην Ευρώπη και να εξετάσουμε πολιτικές και μέτρα. Ποια πράγματα έχουν αποδειχθεί χρήσιμα, ποια διδάγματα ήταν χρήσιμα για την Ευρώπη και πού εντοπίζονται τα σφάλματα. Εν τέλει, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών για την κρισιμότητα των μετάλλων. Όπως είπε η Τζακλίν άλλωστε, ως πολιτικός θα τελούσα εν πλήρη συγχύση. Ποια είναι τα κρίσιμα δηλαδή και όταν θα τα έχουμε εντοπίσει τι θα κάνουμε ώστε να μειωθεί αυτή η κρισιμότητα και ιδίως στην Ευρώπη όπου σε μεγάλο βαθμό είμαστε εξαρτημένοι από τις εισαγωγές των μετάλλων. Ένας τρόπος είναι από τον οργανισμό να γίνουν μελέτες, μεταμελέτες για την αξιολόγηση των δεδομένων που να λάβουν υπόψη και συμπεράσματα και μελετών από τον υπόλοιπο κόσμο και να καταλήξουν σε συμπεράσματα εφαρμογής, δηλαδή για συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί και εδώ ο παράγοντας χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, που μας απευθύνατε το λόγο. Έχω εγγεγραμμένους συναδέλφους. Με πρώτη την κυρία Ρόσπαχ, μετά τον κύριο Αρσένη, μετά τον κύριο Πρόντι, Ντέιβις και ούτω καθεξής. Η κυρία Ρόσπαχ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ειλικρινά με εκπλήσει το εύρος των θεμάτων που πρέπει να καλύψετε. Είναι πάρα πολλά και ποικίλα. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω από τη δικιά μου την πλευρά ποιότητα υδάτων, το ένα. Και το αέριο σχιστόλιθο. Υπάρχουν μελέτες, αναλύσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων μέχρι τώρα. Δεύτερον, μιλάμε για τους... για δοκρινικούς παράγοντες, της τράκτορς. Είναι ένα θέμα που κοιτάτε τι γίνεται με τις καλλιέργειες, δηλαδή γιατί Νομίζαμε ότι από την Βακέλωση, για παράδειγμα, είχαμε απαλληχθεί από άλλους τέτοιους παράγοντες. Αυτά είναι τα θέματα που εμένα με απασχολούν, αλλά επιπλέον θέλω να ρωτήσω κάτι για τις οδικές μεταφορές που μας απασχολεί γιατί αυξάνουν όλο και περισσότερο οι μεταφορές οι οδικές. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις του οξυδίου του αζότου από τι οδικές αυτές μεταφορές. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να κρατήσουμε κάτω από την σημερινή οροφή τα επίπεδα, αλλά τι κάνουμε. Περισσότερες ρυθμίσεις πιστεύετε ότι χρειάζονται ή να βρεθούν άλλοι τρόποι. Και άλλη μια σύντομη ερώτηση. Η ομάδα μου είπε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εισάγουν μια ρύθμιση για όλα τα θεσμικά όργανα έτσι ώστε να υπάρχουν έλεγχοι ε, λογιστικοί. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Ο Κρήτον Αρσένης τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο οργανισμός σας είναι μία από τις υπηρεσίες για τις οποίες, για τις οποίες είμαστε πραγματικά περήφανοι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας οργανισμός ιδιαίτερα ενεργός και τελικά αποδίδει πολύ περισσότερο από όσο αρχικά θα φανταζόμασταν. Και μας βοηθάει όλους το έργο σας. Αυτό που έχω να πω σχετίζονται ακριβώς με αυτό, λοιπόν πάντα για το νομομηθωτικό μου έργο, το δικό μου, χρησιμοποιώ τα δικά σας στοιχεία και ήμουν και μέλος αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου σε Και επειδή πίστευα ότι μπορούν οι ευρωβουλευτές να σας θέτουν ερωτήματα και εσείς να απαντάτε, το έκανα αυτό πολλές φορές για θέματα περιβαλλοντικής σημασίας. Και όντως πήρα απαντήσεις. Πρέπει να το ξέρουν αυτό οι συνάδελφοι και να χρησιμοποιούν αυτή τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός σας. Η Επιτροπή μας θα έπρεπε να φέρει σε πιο στενή επαφή τους ευρωβουλευτές με τον οργανισμό σας. δεν πρέπει το έργο σας να πηγαίνει μόνο στο Προεδρείο ή στους συντονιστές. Πρέπει να φτάνει σε όλους τους ευρωβουλευτές. Εδώ έχω την αίσθηση ότι λείπει ένας κρίκος. Εγώ πριν επισκεφθώ τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, δεν γνώριζα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου σας, αλλά ούτε καν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σχέσης που έχει το δικό σας έργο με τη δικιά μας καθημερινή δουλειά εδώ. Και είναι καλό να ξέρουμε, όπως έμαθα και εγώ τότε, πώς μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε στο δικό μας έργο. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Μακλίντ επίση. πώς βλέπει αυτό το καταπληκτικό έργο, αυτή η φοβερή γνώση, η τέχνη που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει παρετέρω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιήσουν το δικό σας έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αστρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Διευθυντρία για την παρουσίαση που έκανε διεξοδική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι που ξέρει πόση, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει από το Ευρωκοινοβούλιο και για το δικό σας οργανισμό και για την ΕΦΣΑ, διότι η πληροφόρηση αυτή είναι κέρια, ειδικά στους καιρούς μας. Στηρίζω τις προτεραιότητες που εντοπίσατε και προσυπογράφω στις πρώτες, ε, πρώτους στόχους που αναφέρατε για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για τα εδάφη, για την ποιότητα των υδάτων. Ακριβώς ε, αυτό συμβαίνει. Όλο ένα και περισσότερο ανησυχούμε για, τους διαφορετικ... για τις διαφορετικές κατηγορίες ρήπανσης. Υψηλά επίπεδα εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα, χημικά προϊόντα που μπορεί να είναι λιπάσματα, φαρμακευτικά προϊόντα, ε, οσία, ε, οξέα, οτιδήποτε μπορεί να ρυπάνει τα νερά και τη γη μας. Ήθελα λοιπόν να θέσω δύο ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες. Δεδομένου ότι υπάρχει, υπάρχουν όλο και περισσότερο δακτυλίδια τα οποία ανθίστανται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποια μελέτη σχετικά. Διότι έχω λάβει γνώση διαφόρων περιπτώσεων που υπήρξαν οξύτατα περιστατικά ακριβώς λόγω αυτή τη ανθεκτικότητα. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με του θαλάσσιου πόρους. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι και πόσο σημαντική είναι και η διαφύλαξη της θαλάσσια βιοπικιλότητας. Υπάρχουν πρόσφατες έρευνες σε σχέση με την κατάσταση της βιοπικιλότητας στις θάλασσές μας. Για να ολοκληρώσω, να πω ότι Νομίζω καλό θα ήταν να επιδιώκουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους, μακάρι να τους πετύχουμε, αυτούς που έχουμε θέσει για το 2020, διότι βάσει των όσων γνωρίζουμε ότι ήδη συμβαίνουν, θα έλεγα ότι η τάση είναι να επιτεθούν. Αλλά χρησιμοποιείται και ως άλοθη η κρίση για την έλλειψη βούλησης, ιδίως στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Μακλέιντ που είναι μαζί μας. Θα περιοριστώ στο πρόβλημα της προσαρμογής της κλιματικές αλλαγές. Νομίζω ότι είναι κατεπήγη, αυτή η ανάγκη προσαρμογή, αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι ότι ακόμη δεν υπάρχει συνειδητοποίηση αυτή τη ανάγκης. Κάποιες φορές δεν υπάρχει και συνειδητοποίηση των ίδιων των κλιματικών αλλαγών. Λόγου χάρη, ο συσχετισμός με τις γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να γίνεται διότι κάθε τετραγωνικό μέτρο της επικράτειάς μας θα πρέπει να ε, υπόκειται στην ε, λογική της προσαρμογής της κλιματικές αλλαγές. Εάν δεν σκεφτούμε ότι αποτελεί κοινό αγαθό η ασφάλεια της γης μας, της επικράτειάς μας, τότε γενικότερα δεν μπορούμε να δώσουμε θετική διάσταση στη δράση μας και δεν μπορούμε να καταστήσουμε κοινωνούς τους πολίτες αυτής της έννοιας του συλλογικού αγαθού. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα αυτή η έννοια ότι πρέπει να προωθηθεί και να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο από τον οργανισμό σας. Πρέπει να δώσουμε θετική διάσταση ώστε να επιδιώξουμε τους περαιτέρω στόχους μας. Έτσι οι συμπολίτε μας θα έχουν επίγνωση ότι εργάζονται για ένα στόχο και προς όφελος όλων. Θα ξαναπώ τα ίδια που έχω πει και άλλες φορές. Επικοινωνία. Communication. Άφησα την καθηγήτρια Μακλέιτ προσπάθησα να δω τα θέματα λίγο σαν δημοσιογράφος. Άκουσα ιστορίες να διηγείται, άκουσα να μιλεί με τίτλους, όπως σαν διάβαζα τις εφημερίδες. Ασφαλώς αυτά είναι ενδιαφέροντα, αναστατώνουν, άμα τα διαβάζει κανείς, και βοηθούν να φέρουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο κοντά στο περιβάλλον. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Νομίζω όμω ότι ο Οργανισμό Περιβάλλοντο δεν κάνει επαρκή πράγματα για να προωθήσει στη δημοσιότητα το έργο του. Υπάρχουν περιορισμοί για τα όσα πράτεται. Δεν λέω να κάνετε τα πράγματα πιο ελκυστικά. Αλλά ακόμα και οι επιστήμονες και οι φυσικοί κατορθώνουν να βγάζουν τίτλους στα ταμπλόιντ στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας. Δεύτερο, εκτός από τον γενικό τύπο υπάρχουν και πολλοί εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι περιβάλλοντος. Όλοι αυτοί έχουν έρθει να χτυπήσουν την πόρτα σας στην Κοπενχάγη. Έχετε συνεχή επαφή μαζί τους με email. Υπάρχει μια διαρκής ροή ανάμεσα σε εσά και σε αυτούς. Και τέλος, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου λαμβάναμε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού ε, Οργανισμού Περιβάλλοντος. Βέβαια, ομολογώ δεν διάβαζα όλες, διάβασα όμως μερικές. Τώρα δεν παίρνουμε πλέον αντίγραφα, ίσως είναι βέβαια δυνατόν να τα βρει κανείς επιγραμμικά. Αλλά δεν έχω ξαναδιαβάσει καμία από τότε που πάψατε να μου στέλνετε πραγματικά αντίγραφα σε χαρτί. Αυτά. Ο πρόεδρος. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε αν είναι καλύτερα να ερχόμαστε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους για το περιβάλλον με τρόπο που να βλάπτει εν τέλει το περιβάλλον. Κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ καθηγήτρα Μακλέιτ για την παρουσίασή σας. Εγώ μέσα στο iPad έχω όλα τα έγγραφα. Οπότε αυτό με καλύπτει για όλα τα έγγραφα, δεν χρειάζομαι εγώ τίποτα άλλο. Ας διευκρινίσουμε. Μάλλον να ξεκινήσω από το εξή, λέγοντας σας ότι διαπιστώνω πως ε, το τακτικό έργο συνεχίζεται, παρόλο που βάζουμε σε εσά επιπρόσθετα καθήκοντα. Και θέλω να συμφωνήσω και με τον Πρόεδρο και με τον Κρήτον Αρσένη ότι η δικιά μου εμπειρία ως εισηγητής και για την βιοπικιλότητα και για άλλα θέματα ήταν πάρα πολύ θετική. Δηλαδή κάθε φορά που ήρθα σε επαφή μαζί σας πήρα ό,τι βοήθεια χρειάστηκα. Έχω βρεθεί μαζί σας ολόκληρη μέρα και έχω συζητήσει τα διάφορα θέματα. Οπότε είτε ηλεκτρονικά είτε σε χαρτί, διαβάζω τακτικότατα όλες σας τις εκθέσεις. Δεν το αναφέρατε στην παρουσίασή σας μεν, αλλά το διάβασα στο πρόγραμμα εργασίας ότι έχετε και πολλές ε, πολυμερείς δραστηριότητες και μερικές φορές έχω την ε, ε, εντύπωση ότι επιβραδύνεται λιγάκι ο ρυθμός επειδή επικεντρώνεστε στις πολυμερείς δραστηριότητες. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι σημαντικές, αλλά το θέμα είναι μήπως σχεδιάζεται πέρα από τις δυνατότητες που έχει ο οργανισμός. Και τώρα να σας ρωτήσω κάποια πιο λεπτομερή θέματα. Όλοι η ιδέα του να πάψουμε να έχουμε επιδοτήσεις για το περιβάλλον είναι το επόμενο στάδιο, που το επόμενο στάδιο είναι να καθοριστούν οι ορισμοί και η μεθοδολογία. Ίσως θα έπρεπε να είσαστε πιο δραστήριοι και να προκαταλάβετε λίγο τα πράγματα. Τι μπορεί να κάνει, κατά τη γνώμη σας, ο οργανισμός προς αυτή την κατεύθυνση και άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει για την επάρκεια πόρων. Πάντα συζητάμε για δείκτες και για στόχους. Ρωτάω λοιπόν, ο οργανισμός μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και για να βρει τρόπους να θέσει στόχους. Στόχους, ναι. Ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη. Για την χρήση δάτων είναι πολύ δύσκολο να βάλει κανείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ίσως λοιπόν ο δικός σας οργανισμός να μπορεί να μας ε, προσφέρει κάποιο σύστημα για να ε, κάνουμε κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τέλος, Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που άκουσα από την παρουσίαση ότι ο οργανισμός εξακολουθεί να θεωρεί προτεραιότητα την βιοπικιλότητα. Παρ' όλα αυτά εκφράζω ανησυχίε γιατί οι εθνικοί προπολογισμοί μειώνονται βλέπω πίεση για να δίνουν οι χώρες περισσότερη ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την βιοπικιλότητα. Είναι πολύ σημαντικό όμως ο, οργανισμός για το περιβάλλον να επικεντρώνεται στα στοιχεία για την βιοπικιλότητα. Αν χαθούν κάποια είδη, δεν θα τα ανακτήσουμε ποτέ. Γι' αυτό έχετε δίκιο αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν παραπάνω προσπάθειες για την προστασία της βιοπικιλότητας, ίσως καταλήξουμε σε μια κατάσταση η οποία να μην μπορεί πια να αλλάξει καθόλου. Ουλάντα Χίμπνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Χίμπνερ. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ, έχω εντυπωσιαστεί ακούγοντας το εύρος των θεμάτων με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός για το Περιβάλλον. Έχουμε τον Οργανισμό για την Ασφαλεία Τροφίμων, για φάρμακα. Ε, θα λέγει κανείς ότι ασχολούνται με την ποιότητα αυτών των ε, ειδών. Εσείς όμως ασχολείστε με όλα αυτά συγχρόνως. Γι' αυτό και λέω ότι σας θαυμάζω ειλικρινά. Μέχρι τώρα πίστευα ότι επικεντρωνόσασταν μόνο στο περιβάλλον. Ενώ τελικά όλες οι μελέτες που ζητάτε, που αναθέτετε ή που κάνετε εσείς ίδιοι, είναι χρήσιμες και για τη γεωργία και για τη βιομηχανία και για τη δασοκομεία και για την ιατρική, για την έρευνα γενικά. Όπως είπε και ο συνάδελφός σας από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται οι μελέτες σας από όλου. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία για το ποιοι χρησιμοποιούν τις δικές σας μελέτες. Και έπειτα, η βιομηχανία ζητάει τις μελέτες σας. Οι Ινστιτούτα, οι υπηρεσίες ή ακόμα οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών χωρών ενδιαφέρονται, στρέφονται σε εσά για να έχουν πληροφορίες. Κάτι άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, είπατε, για τις κλιματικές αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πλημμύρες, έχουμε ξηρασίες. Έχετε πάρει και προτάσεις από τα κράτη-μέλη, γιατί ξέρετε ποιε περιοχές της Ευρώπης κινδυνεύουν περισσότερο από τέτοια φαινόμενα. Έχετε προτάσεις να τους κάνετε, να τους πείτε «Ε, φτιάξτε δεξαμενέ. ή ξέρω εγώ να φροντίσετε, να βοηθήσετε με στοιχεία. Μόνο δεδομένα συλλέγεται ή κάνετε και προτάσεις στα κράτη-μέλη. Τέλος για την βιοπικιλότητα. Γνωρίζουμε ότι πολλέ χώρες ορίζουν τις περιοχές βιοπικιλότητας βάσει ερευνών. Και μετά από πιο λεπτομερει έρευνες ε, καθορίζονται πιο λεπτομερώς αυτές οι περιοχές ε, βιοπικιλότητας. Πόσο συχνά ε, τα δεδομένα αυτά και απλώς στέλνετε τα πορίσματά σας στις χώρες, υποχρεώνετε τα κράτη-μέλη να σας στέλνουν δεδομένα. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι το εξή. Είπατε 2,5% μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη. Πολύ ευχάριστο να το ακούει αυτό κανείς. Πού οφείλεται στο ότι έχουμε πιο σύγχρονη τεχνολογία που βρίσκει εφαρμογέ στην βιομηχανία ή οφείλεται στο γεγονός ότι η βιομηχανία εγκαταλείπει την Ευρώπη και μεταφέρεται σε άλλα μέρη του κόσμου, στην Ασία για παράδειγμα ή αλλού. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερη επαφή με τους πολίτες. Εσείς προσπαθείτε να αλλάξετε τον τρόπο ζωής των κατοίκων, να αλλάξετε τις συνήθειες των κατοίκων. Μπορείτε να τους δώσετε ξεκάθαρες πληροφορίες. Αν μπορείτε, εμείς μπορούμε να τις προωθήσουμε στις χώρες μας και στους πολίτες μας, αλλά πρέπει να είναι διατυπωμένες πολύ απλά οι ιδέες σας και οι προτάσεις σας για τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στις συνήθειες των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι μόνο μπορούμε να τους τα εξηγήσουμε και εμείς και να τους βοηθήσουμε και όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και με την παραγωγή, με τη βιομηχανία, αλλά έχουν να κάνουν και με την υγεία του πληθυσμού μας. Προσπαθούμε να προωθήσουμε υγιεινούς τρόπους ζωής. Αν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουν οι πολίτες τις συνήθειές τους, συνήθειες διατροφής για παράδειγμα, πρέπει να έχουν σαφή ενημέρωση και απλή. Έρχομαι τώρα στα απορρίμματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε απόβλητα που μεταφέρονται στην Ευρώπη, είναι ένα επιπλέον ε, άχθος που έχει η Ευρώπη. Αλλά δεν έχουμε αρκετή τεχνολογία ώστε να χρησιμοποιούμε τα ανακυκλωμένα απόβλητα. Εσείς έχετε πληροφορίες να μας δώσετε για το κατά πόσο κάπου αλλού στον κόσμο υπάρχουν πιο χρήσιμες, πιο αποτελεσματικές λύσεις. Ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου ανακυκλώνονται μεν τα περισσότερα απόβλητα, αλλά ίσως να μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να έχουμε κάτι καινούριο ώστε τα απόβλητα μετά την ανακύκλωσή τους να καταλήγουν σε κάποια πρώτη ύλη που να μπορεί να χρησιμοποιήσει και πάλι η βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις έθεσαν οι συναδελφοί μου και υπόψη της κυρίας Μακ Γκλέιτ. Θα της δώσω το λόγο για να απαντήσει. Ο κ. Γκερμπράντι αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Είπε όμως ότι οι συνεργάτες του είναι εδώ, θα σημειώσουν ότι λεχθεί. Ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του ή δυνατόν παίρνοντα το τρένο, που είναι λιγότερο επιβαρυντικό για το περιβάλλον, να το πούμε έτσι. Για την κυρία Ρόσπαχ, ευχαριστώ. για το σχιστόλιθο. Λένε ότι ό,τι βρίσκει κανείς κάτω από τον νεροχή του σπιτιού του βρίσκει και στο, ε, στα σχιστολιθικά αέρια. Τώρα, τι να σας πω, εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω κάτι τέτοιο. Ίσως όντως από βάθος, ε, από βάθος να είναι αυσαλέστερη. Δεν είναι βέβαια αποδεδειγμένη η τεχνολογία αυτή. Όμως χρησιμοποιούν χημικά που δεν θα τα ήθελε κανείς να τα βρει στα ύδατα επιφανείας. Είναι λοιπόν μια τεχνολογία η οποία χρειάζεται ένα risk assessment. Για την ώρα δεν διεξάγουμε λεπτομερείς μελέτες. Είναι όμως κάτι το οποίο ανεβαίνει συνεχώς στην ατζέντα μας και ε, πιστεύω ότι ο οργανισμός θα το εξετάσει προσεκτικότερα. Για τα ε, ανθεκτικά μικρόβια δεν έχουμε κάνει καμία συστηματική μελέτη για αυτά. Τώρα για τα μικρόβια στο έδαφος βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχουν φαρμακευτικές βιομηχανίες όπου δημιουργούνται κάποια από τα φάρμακα τα ίδια, το ίδιο το έδαφος ε, είναι γεμάτο από ε, μικροοργανισμούς που είναι ανθεκτικοί. Πρώτη φορά βρέθηκε αυτό ε, στην Κούβα, τώρα το έχουμε δει και στην Ευρώπη μέχρι και σε μια ακτίνα δύο χιλιόμετρων γύρω από τα αρφανακευτικά εργοστάσια. Αν μπει βέβαια στα νερά τότε είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε εμείς ή και οι τρεις οργανισμοί, ΕΦΣΑ και φαρμάκων. Εσείς θα τα αποφασίσετε αυτά για τις οδικές μεταφορές. Δεν υπάρχει βεβαίως θέμα ότι είναι από τα πιο επίγοντα πράγματα που μας απασχολούν σε διάφορες πόλεις και σε διάφορα τμήματα της Ευρώπης προτείνονται πολύ διαφορετικές λύσεις. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι βέβαια ότι η τάση είναι ανωδική. Τώρα το αν έχει σχέση με τις αστικές υποδομές, αυτό πρέπει να αλλάξει είναι η δομή της ζήτησης. Εφόσον επιδοτούνται οι δημόσιες μεταφορές μπορούν να προωθηθούν. Εμείς έχουμε δουλέψει πολύ στον οργανισμό για αυτά. Υπάρχει όμως ένδον αντίσταση. Όταν διαβάζω νέες εκθέσεις από ομάδες που εξετάζουν τις βιώσιμες μεταφορές και ρωτούν μια ολόκληρη γενιά τι αναμένει από τις μεταφορές, βλέπουν πολύ διαφορετικές Ε, διαφορετικά πράγματα. Αυτό που λένε οι λιγότερο από 30 ετών θέλουν δομές, αστικές δομές που θα τους επιτρέπουν να κυκλοφορούν γρήγορα, δεν ενδιαφέρει ούτε αυτοκίνητο να διαθέτουν, ούτε δικό του σπίτι κτλ. Αυτό και εκείνα μπορούν να συναντώνται. Ίσως είναι και θέμα λοιπόν διαφοράς γενεών. Δεν είναι κάτι που θα λύσουμε σήμερα. Δεν είμαι λοιπόν τόσο αισιοδόξη, αλλά υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε με το κοινό και να βελτιώσουμε τις τάσεις αυτές. Αντελήφθη την κωδικοποιημένη ερώτησή σας για τον ΩΣΑ. Η απάντησή μου είναι ότι για τον δικό μας οργανισμό ο ΩΣΑ έρχεται να σπάσει ένα καριδάκι με ένα τεράστιο σφυρί. Υπάρχουν ωστόσο διεθνείς προδιαγραφές που η Ευρώπη μπορεί να έχει την πεποίθηση ότι ευθυγραμμίζεται με αυτές. Και γι' αυτό διερωτώ με αν χρειαζόμαστε κατευθύνες γραμμέ του όσα ή μπορούμε να δούμε τι έχουν και τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλη αυτή η συζήτηση με έχει μπερδέψει λίγο. Έχω διαβάσει με λεπτομέρεια τις guidelines του ΩΣΑ γιατί έχουν βέβαια σημαντική επίπτωση στον οργανισμό μου. Δεν βλέπω να είναι πάρα πολύ ε, σχετικές. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει μια συζήτηση Γι' αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση στην διαθεσμική ομάδα εργασία. Υπάρχουν και άλλε προδιαγραφέ. Και έτσι λοιπόν ανάμεσα αυτέ συζητούνται αυτέ οι άλλε προδιαγραφέ και γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε βέβαια και δεν μπορούμε να σα δώσουμε μια απλή απάντηση ναι ή όχι. Για τον Κρήτονα, ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Και έρχομαι και στην ερώτηση του Κρίς για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε διασυνδέσει και εδώ στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο με τη δική σα Επιτροπή αλλά και με άλλες, πώς να είμαστε πιο παρόντες και παρούσες στην καθημερινή σας εργασία. Αναμένουμε και από εσά να πείτε τι κάνει ο οργανισμό μας. Τώρα θα σας στείλω εγώ αντίγραφα όλες αυτές τις εκθέσεις που έχω εδώ. Hard copies, μην ανησυχείτε, το σημείο σε αυτό που είπατε. Όντως, εμφανιζόμαστε σε τίτλους. Εγώ ήμουνα στην Σαν τελευταία, δίπλα σε μια ομορφωνιά με μπικίνι που δεν ήμουν εγώ βέβαια. Αυτή μιλούσε βέβαια για, την, ε, για τις ε, κρέμες ηλιοθεραπείας, μαυρίσματος. Πάντως εμφανίστηκε ο οργανισμός. Έχουμε και έναν αριθμό ειδικευμένων δημοσιογράφων για περιβαλλοντικά θέματα και βέβαια και αυτοί που ασχολούνται με τα χρηματοπιστωτικά έρχονται στον οργανισμό μας και χρησιμοποιούν το υλικό μας καμιά φορά με λίγες γραμμές, καμιά φορά με παραπομπή στις εκθέσεις μας. Ευχαρίστως να σας καλέσω να κάνετε περισσότερα πράγματα. Κάθε φορά βέβαια που έρχομαι εδώ τα συζητούμε αυτά. Παρ' όλα αυτά, το να απλώσουμε το χέρι, να φτάσουμε κοντά στους πολίτες είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά. Αλλά τα μίντια δεν είναι εύκολος εταίρος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αποφασίζουν τα ίδια τι θα προωθήσουν κάθε μέρα. Και είναι εκπληκτικό το ότι είπαν ότι σήμερα είναι η μέρα της μικρότερης κάλυψης με πάγο της Αρκτικής. Μιλήσαμε στον οργανισμό μας για μια ολόκληρη πενταετία για τις προοπτικές ότι θα μειωθεί η κάλυψη πάγου και ότι πιθανόν δεν θα γίνει αυτό, δηλαδή η ελεύθερη από πάγος αρκτική δεν θα είναι το 2050, αλλά ίσως ήδη το 2020. Πώς καταλήξαμε εμείς είναι βέβαια μιλώντας με ειδικού του ISCAP, με ειδικού ε, δανούς επιστήμονες και ούτε καθεξής. Και κάνοντας και εμείς τις δικές μας μελέτες. Βρισκόμαστε πάντοτε εκεί πίσω από τους τίτλους των εφημερίδων. Καμιά φορά όμως είναι πιο σημαντικό οι επιστήμονες που έχουν κάνει τη δουλειά να εμφανιστούν. Και εμεί τους υποστηρίζουμε βέβαια σε έναν αριθμό ετών για να χρηματοδοτηθούν ε, οι εργασίες τους. Καμιά φορά λοιπόν καθόμαστε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και αυτό ίσως είναι το πρόβλημα. Αν πάτε δηλαδή ένα βήμα πιο κάτω θα δείτε ότι είμαστε εκεί και υποστηρίζουμε αυτούς που βγαίνουν τελικά στους τίτλους. Αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι αποτελεί πρόκληση για όλες και όλους μας να βρούμε κάποια ε, υγιή κοινή λογική και στα όσα κάνουν τα μίδια. για τους endocrine disruptors, αυτά ε, η σχετική μελέτη βεβαίως έφτασε στις, ε, στις σελίδα των εφημερίδων επίσης και στα ψηφιακά μέσα. Μιλήσαμε για τα κύματα καύσωνας, είχαμε ε, πολλούς που ήρθαν στη σελίδα μας, πολύ περισσότερο έρχονται στις ιστοσελίδες μας παρά ε, μέσω των έντυπων μέσων. Τώρα για την με την κατάσταση των ε, επιχειρήσεων που παράγουν ε, οξύδια του άνθρακα. Εμείς συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία, επαγρυπνούμε, το γνωρίζουμε ότι πρέπει να επαγρυπνούμε και βλέπουμε και όλες τις αιτήσει για τη για ε, παροχή δεδομένων από, από εμά. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η γνώση. Εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να έρθουμε στην βιομηχανία και στις χώρες μέλη και να πούμε να αυτά είναι τα δεδομένα σας αλλά να ποια μορφή λαμβάνουν κατά τη δική μας γνώμη. Εμείς και στα δίκτυά μας καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίζουμε ότι η ποιότητα δεδομένων είναι πολύ υψηλή. Κάθε ένα δηλαδή που τα χρησιμοποιεί να μπορεί να βασίζεται σε αυτά. Τώρα, για, την, για τις πληροφορίες, το sharing information, έχουμε διαφορετική άποψη από την ΕΦΣΑ και άλλους οργανισμούς σχετικά με το πώς το ίδιο το περιβάλλον πρέπει να θεωρείται από τους ε, πολίτες ως τμήμα της οικονομίας, όχι ως υποκατάστατο. Η προστασία των φυσικών πόρων δηλαδή είναι το μεγάλο μας μήνυμα. Έχουμε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης με χρήση δηλαδή ε, των πόρων με όχι ληστρικό τρόπο και όχι μόνο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Διότι ένα ελάχιστο ποσοστό των, πόρων, των θαλάσσιων πόρων είναι ακόμα υγιής. Τώρα, η θαλάσσια κοινότητα στο σύνολό της βλέπει δύο τρόπους. Αφενός με marine protected πάρα πολύ σημαντικό, χώρος προστατευόμενος δηλαδή στη θάλασσα και εν της αλλαγής του κλίματος, όπου βλέπουμε ότι ορισμένοι από τους σπόρους έχουν μετακινηθεί, βρίσκονται σε άλλες τοποθεσίες από ό,τι ήταν πριν, αλλά ταυτόχρονα και για την τεχνολογία ε, που έχει σχέση με τα φύκια, τη βιοενέργεια και άλλα σχετικά. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα νέα, θα τα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, θα βρείτε και τη βιοπικιλότητα και όλοι αυτή την έρευνα που γίνεται για τα απορρίμματα, για τους σημαντικούς προστατευόμενους χώρους στη θάλασσα, θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών, παρουσιασμένο με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο από τους ίδιους τους ερευνητές. Για τους στόχους τώρα. Πολύ σύντομα. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα στόχων και όταν μας ρώτησε μια ομάδα ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή μας πέρα από τα χημικά στο περιβάλλον είναι πώς να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι στόχοι που έχουμε στα λεγόμενα flagship κτλ δεν άλληλο ακυρώνονται. Για παράδειγμα, οι στόχοι της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της κοινή αγροτικής πολιτικής, της κοινή πολιτικής αλίας και άλλων τμήματων της οικονομίας να μην αρχίσουν να υποσκάπτουν οι μεν του δε. Και γι' αυτό επανέρχομαι στην ιδέα του Natural Capital Accounting, τη καταγραφή ε, της καταγραφής των φυσικών κεφαλαίων. Και μέσα στο εξάμεινο είναι δυνατόν να γίνει μια ε, γνήσια αξιολόγηση για το πώς, το χρησιμοποιείται ένα μέρος της βάσης για να ενισχυθεί άλλο μέρος της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη ε, να επιλέξει μια πολύ υψηλή ποιότητας ε, λογιστική προσέγγιση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για άδειε χρυσή άδειε εξόριξη κτλ. Γιατί χωρίς τις βάσεις αυτές δεν μπορούμε παρά να μείνουμε στο περιγραφικό επίπεδο και έτσι δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις. Για την αλλαγή του κλίματος και την προστασία της κοινή μα κληρονομία, επανέρχομαι στο ότι ο μόνος τρόπος είναι να εξηγήσουμε καλύτερα και στο κοινό και στα θεσμικά όργανα. Και ένας παράγοντας είναι να δούμε πόσο απομονωμένες είναι πολλές διοικητικές αρχές από τη συζήτηση που γίνεται εδώ. Ήμουνα στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα και διαπίστωσα ότι μια από τις αυτόνομες περιφέρειες που δείχνει πραγματικά πάθος για να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά δίκτυα και με τους πολίτες που επιθυμούν να μπουν σε θέματα βιοπικιλότητα κτλ. Υπήρχε δηλαδή πραγματικά αυτή η επιθυμία ανάμεσα σε αυτά που βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν και θεωρούν ότι δεν έχουν ακόμα διασυνδεθεί αρκετά με την προσπάθεια να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια λοιπόν με τις τοπικές ε, ε, δημόσιες αρχές για να δούμε τι μπορούν να κάνουν και όλα αυτά να διασυνδεθούν με την προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων. Γιατί αυτοί οι στόχοι δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν από το τίποτα. Χρειάζεται να συνεργαστούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και εδώ επανερχόμαστε βέβαια στην επικοινωνία και τη βελτίωσή της. Μπορούμε να δώσουμε συμβουλές, όπως ανεκάλυψε ο Κρήτον, αν με πάρετε τηλέφωνο θα σας δώσουμε πληροφορίες. Όσο περισσότερες μπορούμε μάλιστα στη βάση των πόρων που διαθέτουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συνεργασία μας δήμους και κοινότητες σε ένα επίπεδο είναι απόλυτα σημαντική για να εξασφαλίσουμε ότι οι ε, ε, πληροφορίες που θα έχουμε θα παίξουν το ρόλο του καταλήτη για να αναλυφθεί δράση. Βεβαίως υπάρχει επικουρικότητα, έτσι δεν είναι, και χρειάζεται να την τηρούμε. Παρ' όλα αυτά, κάτι που θα θέλαμε να θεωρηθεί ο οργανισμός μας είναι ως καταλήτης για να προσφερθεί μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών παροχής συμβουλών που να μπορέσει πραγματικά να μεταφραστεί η γνώση που έχουμε σε τοπική δράση. Πραγματικά, πάνω-πάνω στο κατάλογο πρέπει να βρίσκεται η εφαρμογή. Έχουμε στέρεα νομοθεσία. Αν εφαρμοστεί σωστά θα αλλάξει πολλά πράγματα επί τόπου. Πολλές τοπικές αρχές δεν είναι διασυνδεμένες με πολλές από τις βέλτιστες πρακτικές και αυτό είναι δική μας δουλειά αλλά και καθενός δουλειά να το καταστήσει αυτό γνωστότερο. Επομένως, συμβουλές που δίνονται σε τοπικό πλέον επίπεδο. Αυτό είναι ασφαλώς απαραίτητο ε, τμήμα του πακέτου. Είτε πρόκειται για παροχή συμβουλών και πληροφοριών σε μικρές ε, επιχειρήσεις ή σε μεγαλύτερες βιομηχανίες για να κάνουν αυτά που μπορούν και που λένε στις δημόσιες σχέσεις τους και βεβαίως συμμετοχή των πολιτών είτε σε επιστημονικά προγράμματα και βέβαια και εν ώψη της τεράστιας ανεργίας. Είχαμε μια προσφορά από την Ισπανία να μπουν ένα μέρος των ανέργων σε προγράμματα πολιτών προστασίας της βιοποικιλότητας. Αυτά είναι σημαντικά για να δοθεί και μια θετική εντύπωση στον κόσμο πώς μπορεί το περιβάλλον να παίξει ένα θετικό ρόλο στην ανάπτυξη και να δημιουργηθούν και αυτές οι 400.000 θέσεις απασχόλησης που ανέφερε πριν ο Πρόεδρος σας. Ευχαριστώ για την πλήρη απάντηση των ερωτήσεων που έδειξε για μια ακόμη φορά ότι στην Κοπενχάγη ο, ο οργανισμός περιβάλλοντος έχει πραγματικά σημαντική γνώση και επιθυμία να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο. Επίσης, επισημαίνω ότι ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος, ας μην το λησμονούμε αυτό, και αυτό, σε αυτό αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και ο οργανισμός αλλά και όλοι οι οργανισμοί και για μας ως κοινοβουλευτικούς είναι σημαντικό να μπορούμε να πούμε ότι εν τέλει διότι μιλούμε πολύ για χρήματα και πού επενδύονται τα χρήματα. Με τους οργανισμούς μας, στην ουσία, εξοικονομούμε σημαντικά κονδύλια. Δεν χρειάζεται μια δουλειά να γίνεται 27, 27 φορές, σε 27 χώρες δηλαδή. Ο οργανισμός σας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για δημοτικές αρχές, για ομόσπονδα κρατήδια, για χώρες μέλη και ούτε Σας ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εργασία σας με θετικό κριτικό πνεύμα, αυτό είναι σαφές, και σας εύχομαι καλή επιτυχία και όπως είπα θα παρακολουθούμε την εργασία σας κριτική αλλά με δίκαιο και ανθρώπινο τρόπο. Αποδίδω πολύ μεγάλη αξία σε αυτό και νομίζω ότι και όλοι οι συνάδελφοί μας που ήταν παρόντες και παρούσες δεν ήταν πολύ μεν, αλλά όσοι ήταν παρόντες παρακολούθησαν πολύ προσεκτικά τα όσα δημιούργησαν εδώ και μας ενδιέφεραν πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά από σας σήμερα και ήταν πραγματικά το απόγευμά μας πλήρες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διάταξής μας. Ευχαριστώ όλες και όλους που ήρθαν και επίσης και τους συναδέλφους του Management Board. Ευχαριστώ πολύ. Λίγη η συνεδρίαση και η επομένη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Καλή επάνωδο στις αιστείες σας.